Okay, colleagues. Um, this is our last vote before the Easter break, so we have. Συνάδελφοι, να ψηφίσουμε πριν την ε, τελευταία ψηφοφορία πριν το Πάσχα. Ε, δύο συζητήσει, η μία για την Αφρική, η άλλη για τα φορολογικά, αλλά κάνουμε πρώτα τι ψηφοφορίε μα. Να κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο υπέρ παρακαλώ του να κάνουμε τα υποπέσει για το Πάσχα. Τώρα να ψηφίσουμε.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 So, okay, the... Μάλιστα, πέρα ψηφοφορία. 17 ψήφοι, 15 υπέρ. Δύο εποχέ όσοι απήχαν να μην πάνε διακοπέ για το Πάσχα. 17 λοιπόν άτομα, εντάξει, ψήφισαν όλοι πολύ ωραία. Τώρα να σοβρευτούμε λίγο. Ψηφίσαμε στους συντονιστές για τις προφορικές ερωτήσεις για τα ODAs, επίσημη αυτοξιακή βοήθεια. Τώρα λοιπόν ε, να ψηφίσουμε τις ερωτήσεις για την Επιτροπή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. The vote is closed. Πέρα ψηφορία. 15 υπέρ, ένας κατά καμία αποχή. Ευχαριστώ, εγκρίθηκε αυτή η ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση η ίδια ουσιαστικά ερώτηση, αλλά προ το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Ευχαριστώ και τώρα λοιπόν αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε στην Ολομέλεια του Απριλίου. Αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι πολιτικέ ομάδε για να το πετύχουν αυτό. Και τώρα περνάμε στην τρίτη ψηφοφορία. Πρόκειται για ένα διορθωτικό, πολύ μικρό διορθωτικό, για το ε, εθελούσιο Ευρωπαϊκό Σώμα. Ένα ψηφοφορία. Πέρασε. 16 υπέρ κανεί κατά μία αποχή. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνονται, ολοκληρώνονται λοιπόν οι ψηφοφορίες μας. So we can move on now to item 17. Περνάμε λοιπόν στο 17. Ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκτησης για τη Συμφωνία για το Εμπόριο, την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να λεφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας. Έρχεται το σχέδιο έκθεσης, δεν έχουμε λάβει τροπολογίες και ο κύριος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, είναι τεχνικό το ζήτημα. Είχε γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η Κροατία προσχώρησε στην Ένωση τον Ιούλιο του 2013 και γι' αυτό λοιπόν ε, προτείνεται ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία με την ε, Νοτιοφρική για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αρχικό πρωτόκολλο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και από την Νότια Αφρική το Δεκέμβριο του 2014, αλλά η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση θέλει να αποφασίσει τώρα την υπογραφή του πρόσθετου πρωτοκόλου. Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχουν νέε εξελίξεις ως προς αυτή την υπόθεση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία για την εκδήλωση την τέλετη υπογραφής. Αυτό δεν αποτρέπει φυσικά να ψηφίσει η Επιτροπή μας, αλλά πριν την υπογραφή δεν μπορούμε να έχουμε την τελική συνένεση από πλευρά τη Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο. Ο κύριο Λίτ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Στυρ για την εργασία του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Σα ευχαριστούμε όμω για την εργασία σα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν είναι το κανεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση που θέλει να πάρει το λόγο. Νομίζω ότι είναι μάλλον τυποποιημένη αυτή η διαδικασία. Θα συνεργαστούμε με την ε, γραμματεία, λέει ο κ. Στήρ. Θα θέλαμε να ξέρουμε την ημερομηνία της τέλετης υπογραφής, αλλά αυτά συνοηθούμε αυτά με την γραμματεία για να ξέρουμε και για την ακριβή ημερομηνία για την Επιτροπή. Τον Απρίλιο κατά πάσα πιθανότητα λέει η Πρόεδρος. Ωραία, περνάμε λοιπόν στο 14. Το δικαίωμα στο νερό. Η συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Θα ξέρετε ότι συγκεντρώθηκαν ένα εκατομμύριο υπογραφές για να υπάρξει μια πρωτοβουλία των πολιτών Δικαίωμα στο νερό. Έχουμε μία γνωμοδότηση του κυρίου Πρέντα για το θέμα αυτό. Να δώσουμε λοιπόν στον κύριο Πρέντα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φαντάζομαι έχετε λάβει το κείμενο της γνωμοδότησης με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2015. Δεν ναι, είναι και μακροσκελές. Είναι ένα σύντομο κείμενο και τώρα θα προσπαθήσω να το συμπληρώσω με ορισμένες προφορικές παρατηρήσεις γενικού χαρακτήρα. Καταρχάς γνωρίζετε ότι αυτό που εμείς ότι είναι πολύ φυσιολογικό και απλό, δηλαδή το να ανοίγουμε τη βρύση, δεν είναι το ίδιο αυτονόητο σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. Εδώ έχουμε κάποια διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία βέβαια δεν είναι και πάντοτε εντελώς αξιόπιστα. Θεωρούμε όμως ότι είναι αξιόπιστες εκτιμήσεις. Τα 748 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο νερό και δεν έχει τη βασική αποχέτευση το 1 τρίτο. 4.000 παιδιά δε φαίνεται ότι πεθαίνουν καθημερινά λόγω ασθενειών που οφείλονται ε, είτε στην έλλειψη νερού, είτε σε μόλυνση του νερού και στην κακή υγιεινή. Έχουμε πολλά στοιχεία για θανάτους ε, βρεφών ε, κάτω των 5 μηνών που πεθαίνουν καθημερινά από διάρρεια. Και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι αριθμοί μας δίνουν μία εικόνα που κατέμασε ένα είναι Βέβαια, έχει αναλυφθεί η δέσμευση πλέον για να υπάρξει πρόοδο σε την πρόσβαση στο νερό, στο καθαρό νερό και στην ε, εξυγίανση και στις υπηρεσίες και αποχέτευσης για να έχουμε μια ζωή αξιοπρεπή και υγιή για όλους. Η δική μας επιτροπή που γνωμοδοτεί, αρμόδια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, θέλουμε να περιλάβουμε την βελτίωση της πρόσβασης στο νερό, την εξηγένση. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται συζητήσεις Υπάρχει και διάσταση του φύλου, γιατί σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες είναι αυτές που παραδοσιακά είναι υπεύθυνε με τον κύριο Νόιζερ πριν από κάποιες εβδομάδες και με το φίλο Κορά εδώ πέρα, το φίλο μου, ήμασταν στο Τατζικιστάν. Euh, euh. Και είδαμε γυναίκες να μεταφέρουν ε, νερό με μεγάλα μπιντόνια. Δεν ξέρω πού το βλέπουμε αυτό ακόμη στις μέρες μας. Υπάρχει και αυτή η διάσταση. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες στον τομέα υγιεινής αποχέτευσης ίδρυυσης, WASH, 1,5 δις ευρώ ετησίως. Σημαντικό το ποσό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, διότι πολύ συχνά αυτοστιγματιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο, λησμονώντας ότι η προσπάθεια που καταβάλουμε παρόλα αυτά αξιοσημείωτη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, να ασκούμε ανόητη κριτική, ανόητη αυτοκριτική. 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύουμε τις ίδιες τις χώρες για όλα αυτά όπως έδειξε και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου του 12, μπορούμε ακόμη να βελτιώσουμε περισσότερο αποτελεσματικότητα. Πάντοτε επιδέχεται βέβαια βελτιώσει κατάσταση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ουσιώδη και είναι σημαντική η συνεισφορά μας. Τώρα προτείνω επίσης ορισμένε λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης εντός του δικού μας πεδίου αρμοδιοτήτων. Πρώτα απ' όλα θέλουμε η διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή ε, ότι πρόσβαση στο νερό, πόσιμο νερό, καθαρό νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Επίσης πρέπει να στηρίξουμε τη συμπερίληψη ενός στόχου για την ε, βιώσιμη διαχείριση του νερού, την υγιεινή για όλους μέχρι το 2030 στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για μετά το 2015. Το Σεπτέμβριο θα τα αποφασίσουμε αυτά. Στην παράγραφο 2 της ε, γνωμοδοτησής μου το λέω αυτό. Επίσης λέω ότι θα πρέπει να ψηφίσει και εθνικοί υπερπολογισμοί να εστιάσουν περισσότερο στον τομέα ΟΑΣ. Σα είπα τι σημαίνει αυτό το ακρονίμιο. Νερό, ίδρυψη, αποχέτευση, υγιεινή. Διακυβέρνηση διαχείριση νερού, ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε ανισόμενε χώρε, λαμβάνοντα υπόψη τι ανάγκε ε, του ευάλωτου πληθυσμού, ιδίω στην Ήπεθρο. Θα πρότεινα επίσης ότι πρέπει να στηριχθούν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης όπως το Global Water Solidarity Platform, πρόγραμμα των νόμων για την ανάπτυξη, μηχανισμοί του είδους 1% αλληλεγγύη για το νερό και την αποχέτευση, ίδρυυση αποχέτευση. Το έχω βάλει και αυτό και για αυτή τη στρατική μα μετά το 2015 λέω ότι πρέπει να έχουμε έναν παγκόσμιο μηχανισμό παρακολούθηση και ελέγχου για να βλέπουμε τι πρόοδο συντελείται σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε καθαρό νερό και στη διαχείριση του νερό βιώσιμου πόρου. Στη γνωμοδότησή μου αναγκάστηκα βέβαια να περιοριστώ γιατί υπάρχουν δρακόντια μέτρα, ε, δρακόντιοι περιορισμοί για τη μετάφραση. Άρα δεν έπρεπε να μακρηγορήσω, ε, χρειάστηκε να τροποποιήσω τη γνωμοδότησή μου για να κόψω κάποια και να αναπτύξω καλύτερα τα βασικά σημεία. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Um, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο, η Μαρία Χόλμπρουκ. Α, Έλλη Σλάιν πρώτα. Η Μαρία. Πρώτα η Μαρία και η Έλλη εν συνεχεία και ο Ιγνάθιο θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Το Νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι θα ήθελα να το εκφράσω, γιατί πρόκειται για μια απαραίτητη προϋπόθεση για να επιβιώσει κανείς. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει. Ξέρουμε ότι είναι άδικη η πρόσβαση στο νερό δεν μπορούμε να πούμε ότι πλήττεται ιδιαίτερα η Ποσαχάρια Αφρική, η χύψη χώρα. Η έκθεση της ΠΟΗ και της UNICEF καταδεικνύουν ότι υπάρχει βελτίωση, αλλά υπάρχει ανισότητα. Και ιδιαίτερα μειονεκτούντες είναι οι περιοχές της υπαίθρου σε σχέση με τις αστικές περιοχές και φυσικά υπάρχει και μεγάλη αστική διαφορά. Οι φτωχοί έχουν πολύ πιο δύσκολη πρόσβαση στο πόσιμο νερό από ότι οι πλούσιοι. Και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί τώρα στην έκθεση. Για τη χρηματοδότηση είπατε δύο λόγια. Όταν μιλάμε για χρηματοδότηση της παροχής νερού, πρέπει να κοιτάξουμε το κατά πόσο χρειάζομαστε δημόσια υδροδότηση ή κατά πόσον θέλουμε να γίνει ιδιωτική υδροδότηση. Εγώ θεωρώ ότι αποτελεί δημόσιο αυτό το νερό και θα πρέπει να παραμείνει στα δημόσια χέρια. Υπάρχουν όλο και πιο πολλέ συμπράξεις ε, ε, δημοσίου και δημοσίου τομέα των διαφόρων περιοχών δηλαδή και περιφερειών. Αν υπάρξει ιδιωτικοποίηση θα έχουμε πολλά αρνητικά παραδείγματα και αυτό που φαίνεται με τον όμιλο Νεσλέ που εκμεταλλεύεται την κατάσταση, γεμίζει με νερό μπουκάλα και τα πουλάει πανάκριβα σε περιοχές που ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ζήσει. Θα πρέπει το πόσιμο είδωρ να διατίθεται σε όλους. Στην Ιγυρία Νομίζω το νερό είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη. Νομίζω ότι κάτι κάνουμε λάθο. <coughs> Δεν ε, πετυχαίνουμε του στόχου μα. Δεν μπορεί να είναι το μέλλον αυτό. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει κάπου στην έκθεση. Um, um, Ευχαριστώ. Άλλη Λάινεκ, εκ μέρου της Πατρίτσια Τόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σκιώδη εισηγήτρια Πατρίτσια Τόγια δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ και γι' αυτό έχω ένα σημείωμα που πρέπει να σα διαβάσω εξ ονόματό τη. Ευχαριστώ τον εισηγητή Βαν Μπρέντα για την καλή του εργασία. Ωστόσο, δυστυχώ το νερό σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι θέμα προτεραιότητα και εμεί οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε θέμα προτεραιότητα. Ωστόσο, αποτελεί ένα πολύ λεπτό θέμα που αποτελεί και αίτιο συγκρούση. Είναι σημαντικό για, για τομεί όπω αυτή τη ενέργεια ή γεωργία επόμενη, στην επόμενη σύνοδο για τις κλιματικές αλλαγές το θέμα του νερού θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Για να εστιάσουμε στη σημερινή προσοχή θεωρώ πως ένα τέτοιο θέμα όπως η πρωτοβουλία από το πολιτών θα έπρεπε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Αυτή η γνωμοδότηση μαζί με τη συζήτηση στην Επιτροπή ΕΜΗ θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για να τονιστεί η σημασία του θέματος και να ε, ξεκινήσει και πάλι με νέα όθηση η πρωτοβουλία των πολιτών. Πρόκειται για ένα κοινό αγαθό που ποτέ δεν μπορεί να αποτελέσει ένα εμπόρευμα. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το στόχο να αγγιθούμε για όλους μέχρι το 2030 πόσιμο νερό και ε, κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Η πρωτοβουλία για την αλληλεγγύη για το νερό και για τις υπηρεσίες της υγιεινής θα πρέπει να είναι ε, μια πρωτοβουλία που θα στριχθεί από όλους. Επίσης θα πρέπει να έχουμε στόχο τη δημιουργία και τη βελτίωση των υποδομών που στόχο έχουν την υδροδότηση σε πόσιμο νερό και τα βασικά, ε, τις βασικές υγειονομικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Ο Νιάτζιο Κοράου. Σας ευχαριστώ. Εγώ βασικά συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος Πρέντα. Μάλιστα παίρνω λαδί από τον προβληματισμό που κάναμε στο Τατζικιστάν όταν είδαμε τις γυναίκες να κουβαλάνε τα μπιτόνια με το νερό. Ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στο Τατζικιστάν είναι ότι οι πηγές που προέρχονται, που ξεκινάνε από το Ουσβεκιστάν, δεν μπορούσαν τελικά να φτάσουν για να πάνε σε, όλα τα χωριά γιατί το νερό χρησιμοποιούταν ε, για την εντατική ε, καλλιέργεια βαμβακιού η οποία ελέγχεται από τις τεράστιες κινέζικες ε, πολυεθνικές. Πιθανότατα, μένοντας στο θέμα της αναπτυξιακής πολιτικής, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε στις υποδομές που φέρνουν την υδροδότηση στα χωριά και στις πόλεις να είναι μια προτεραιότητα και να μένουν στο δημόσιο τομέα. Γιατί όπως έλεγε η συνάδελφος όπως ένα μεγάλος κίνδυνος είναι να θεθεί η διαχείριση του νερού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός στα χέρια των ιδιωτών. Γιατί όταν είναι θέμα κέρδους είναι λογικό ότι η υπηρεσία αυτή θα είναι προβληματική. Εμείς είμαστε υπέρ του να θεωρηθεί το νερό ως ένα ανθρώπινο δικαίωμα και η πρόσβαση στο νερό. Δυστυχώς όμως ακόμα και σήμερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει παντού ελεύθερη πρόσβαση στο νερό και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο νερό. Κυρία Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σας εκφράσω τις σκέψεις μου γιατί είναι εξαιρετική κατά με δουλειά του κυρίου Πρέντα. Αλλά και έχοντας υπόψη μου άλλες επιτροπές, ε, παραδείγματο χάρη, ε, την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών, η μόνη που είχε επιτυχία, είναι κάτι που μας είχε απασχολήσει και ιδίως αυτή τη στιγμή που επίκειται αναθεώρηση του κανονισμού περί ε, πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών που είναι το βασικό εργαλείο της συμμετοχής των πολιτών και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή είναι η μόνη, όπως είπα, σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την ε, περίοδο προβληματισμού για την αναθεώρηση αυτού του κανονισμού Μία από τις πτυχές ε, που από την Επιτροπή Αναφορών, γιατί σε αυτή την Επιτροπή αναφερόμουν και επειδή είμαι εισηγήτρια, εκεί θα θέλαμε η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών να μπορεί να προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στις συνθήκες που θα άπτονται συγκεκριμένων ζητημάτων. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, Είμαστε πεπισμένοι όλοι για το κατά πόσο είναι δικαίωμα ή όχι το νερό ο ΙΕ, οργά, ε, συγγνώμη, πριν από πέντε χρόνια το είπε ξεκάθαρα και για την ε, ε, αποχέτευση και για το καθαρό πόσιμο νερό που όχι είναι απλά ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απαραίτητα, ε, είναι προϋποθέσεις και για να μπορούν να είναι εξασφαλισμένα και τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη έχουν υποχρεώσεις για την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης αυτό το νερό να είναι προσβάσιμο, να είναι ε, κατάλληλο και εμείς ε, Έχουμε και το άρθρο 208 της συνθήκης όπου ορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους ε, της αναπτυξιακής ενεργασίας για την εφαρμογή των πολιτικών που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες και μια πολιτική είναι να έχει μεγαλύτερη συνέπεια και συνεκτικότητα η πολιτική μας. Έχουμε την αρχή των ε, Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε. Όπως ήδη είπαν οι συνάδελφοι, το νερό δεν είναι ένα απλό προϊόν. Η οδηγία 2060 λέει ότι δεν είναι εμπορικό αγαθό, είναι κληρονομιά το νερό και τελικά δεν είναι το θέμα να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Σε καμία περίπτωση Ήδη έχει δρομολογήσει πρωτοβουλίε η Ένωση για να επαγρυπνήσει και να φροντίσει ότι θα έχουν οι Ευρωπαίοι ε, το δικαίωμα στη, στο νερό και στην αποχέτευση, θα μπορούν να το ασκήσουν. Αυτό είναι, αναφέρει το δικαίωμα, δεν τίθεται από αμφισβήτηση. Είπαμε ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερο χρηματοδότη. Μέσω του προγράμματο Water Supply, Sanitation και Hygiene θα μπορούσαμε να δράσουμε περισσότερο πάνω στο τομέα αυτό. Και ένα από τα σημαντικά στοιχεία του σχεδίου γνωμοδότηση του κυρίου Πρέντα είναι το ότι επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι ένα από του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, η πρόσβαση στο νερό δηλαδή και την αποχέτευση, και συμφωνώ βέβαια, ε, δεν θα πρέπει επίσης όμως να μας διαφεύγει το ότι θα πρέπει να ε, μπορούμε να συμμετάσχουμε όχι μόνο σε αυτό το στόχο αλλά και στην, ε, στον καθορισμό των στόχων και των δικτών για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτόν τον την παρακολούθηση. Στία. Ο κύριος Στία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα, δηλαδή και από την οπτική γωνία των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015 και ιδίω το στόχο 6, διαθεσιμότητα και βιώσιμη διαχείριση του νερού και της ε, αποχέτευσης. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό και σε όλες τις γνωμοδοτήσεις μας πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε αυτό το πλαίσιο των νέων στόχων του νέου αναπτυξιακού πλαισίου. Πιο γενικά τώρα, <clears throat> χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει σοβαρά αυτή την πρωτοβουλία, όπως δεν συνέβη με προηγούμενες. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. the last speaker. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν έχει κάτι να πει. Δεν γνωρίζω τα ονόματά σας. Ονομάζομαι Πολ Τσικαρέλη και εργάζομαι στην DigiDevco και είμαι τμήματάρχης για το νερό, του τμήματος για το νερό. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την ε, ε, δέσμευση και προσήλωση της Επιτροπής στο θέμα του νερού και ε, των υγειονομικών υπηρεσιών από το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο όπου δώσαμε ε, πρόσβαση στο νερό σε 75 εκατομμύρια ανθρώπους και ε, υγειονομικές υπηρεσίες σε άλλα τόσα. Πολύ μεγάλα νούμερα δηλαδή. Με το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ατζέντα για την αλλαγή, το νερό δεν θεωρείται μόνο ως ε, νερό και υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και ως ένα ε, ε, ε, οριζόντιο ζήτημα και γι' αυτό δουλεύουμε και στην διασυνοριακή διαχείριση του νερού καθώς και σε σχέση με τη σύνδεση ανάμεσα στο νερό, την ενέργεια και την ασφάλεια στα τρόφιμα. Και αυτό γιατί όπως υπόθηκε και από κάποιους ευρωβουλευτές βλέπουμε ότι συχνά υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στη χρήση του νερού σε, το, σε περιοχές όπου για παράδειγμα υπάρχει πολύ μεγάλη χρήση του νερού για τη γεωργία εις βάρος των ανθρώπων που δεν έχουν ε, καν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης θέλω να σας πω ότι η Κομισιόν αναπτύσσει ένα, μια εργαλειοθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου ε, σχεδόν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, ε, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε και να δούμε πώς ε, διαχειρίζεται την ανθρώπινη συνιστόσα το πρόγραμμα. Αυτό θα μας ε, διαβεβαιώσει ότι δίνεται έντονη ε, προσοχή στο θέμα της πρόσβασης στο νερό. Το θέμα τώρα της ε, εταιρική σχέσης μεταξύ δημόσιου και δημόσιου, η Κομισιόν ε, πιέζει όχι μόνο για τη ε, δημόσια-δημόσια εταιρική σχέση, αλλά και για δημόσια-ιδιωτική εταιρική σχέση. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι βλέπουμε το νερό σαν κέρδος, κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά μόνο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούμε ότι ο ιδιωτικό τομέας μπορεί να είναι ο πάροχος της υπηρεσίας ενώ οι υποδομές παραμένουν δημόσιες. Ο βασικός στόχος που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι η καθολική πρόσβαση στο νερό, προσιτό, βιώσιμο και καθολικό τρόπο. Δηλαδή νερό για όλους, αλλά μέσα σε ένα σύστημα το οποίο να είναι βιώσιμο. Και αυτό κάποιες φορές απαιτεί την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με ότι υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο που ε, ενισχύει και ότι η πρόσβαση στο νερό θα είναι εγγυημένη ακόμα και για τους φτωχότερους των φτωχών. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και αριθμητικά στοιχεία, αλλά κανονικά εδώ έχω ολοκληρώσει την ε, παρέμβασή μου. εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέντα, έχετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τον εκπρόσωπο της ΔΕΦΚΟ που μας ε, μίλησε. Κάποια σημεία που αποτέλεσαν αντικείμενο των παρεμβάσεων ήδη είναι η ουσία των τροπολογιών που έχω συντάξει, γιατί όπως σας είπα χρειάστηκε να, μειώθει, να το κείμενο, να γίνει πιο σύντομο. Οπότε προβλέψαμε τροπολογίες που θα το συμπληρώσουν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις προτάσεις σας και ελπίζω ότι θα μπορέσω να χαίρω τη στήριξη διαφόρων πολιτικών ομάδων. Τώρα βέβαια υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε, να μην μπούμε τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες. Θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε ε, επί τη βάση των τροπολογιών. Πάντως, ε, γενικά, θέλω να πω ότι πρέπει να εστιαστούμε εδώ στην πτυχή της ανάπτυξης, για την γνωμοδότηση που κάνουμε εμείς ως ε, Επιτροπή για την Ανάπτυξη προς την ΕΝΒΗ. Δεν είναι νομίζω αυτός ο χώρος. Τώρα η φίλη Γερμανίδα με συζητά με την κυρία Χάουτα, αλλά θα το πω παρόλα αυτά, ότι η ιδέα δηλαδή είναι ότι εδώ δεν χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις ιδεολογικές μας διαφορές ε, με τις πολυεθνικές. Είναι κρίμα που συζητούν. Κυρία αλλά Χάιδη, θέλω να πω κάτι για εκείνην. Ναι. Έλεγα λοιπόν πως ίσως είναι χρήσιμο για το δικηπολιτικό μας διάλογο. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να εστιαστούμε στην γνωμοδότηση ως γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης για τους συναδέλφους της Επιτροπής ΕΝΒΗ και ίσως να μην είναι ο κατάλληλος χώρος για να ρυθμίσουμε τις διαφορές μας και τις ιδεολογικές μας διαφορές την τοποθέτηση των διαφόρων ε, ομάδων σε σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία ή τον καπιταλισμό. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση που προέρχεται από την πλευρά της αναπτυξιακή και αφορά την πρόσβαση στο νερό. Δεν είναι εδώ όμως ο χώρος για να ορίσουμε το καθεστώς των ε, πρωτοβουλειών των πολιτών. Αυτό είναι θέμα που απασχολεί την Επιτροπή ΑΦΚΟ, της οποίας είμαι μέρος, μέλος. Ε, πρέπει να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς, δηλαδή να ε, αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ και άρα ε, έτσι να ε, συντάξουμε και τη γνωμοδότησή μας. Δεν θα ρυθμίσουμε δηλαδή εδώ όλες τις παγκόσμιες συγκρούσεις και τις ιδεολογικές διαφορές. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της πρόσβασης στο νερό Αυτή, αυτό πρέπει να είναι το φόρμα, το φόρμα, τη μορφή, Η διαφορετικά θα είναι πολύ ε, μακρύ ο σκελές το κείμενο, θα τα βάλουμε όλα και κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Βουσκό έφτασε και το τελευταίο σημείο. Σκοπεύουμε να το μεταφέρουμε. Θα το συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε την ατζέντα έτσι όπως είχαμε προγραμματίσει αρχικά, αν συμφωνεί και η κυρία Χόλμπρουκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προθεσμία για τροπολογίες είναι η μεθεπόμενη εβδομάδα, 14 Απριλίου, για την δομοδότηση του κυρίου Πρέντα. ψηφίζουμε 6 Μαΐου. Για την γνωμοδότηση αυτή. Συνάδελφοι, μας περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το 15. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Και χαίρομαι που μαζί μας σήμερα έχουμε τον Νίκ Βέσκοτ, ο οποίος είναι Διευθυντή τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για τα θέματα Αφρική επέστρεψε μόλι από την Ιγυρία όπου έχουμε μια ιστορική αλλαγή τη πολιτική ε, εξουσία μετά τι εκλογέ. Πείτε μα και λόγια και για πολλά άλλα ζητήματα. Οι συντονιστέ τη Επιτροπή μα θεώρησαν ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να εξετάσει η Επιτροπή μα ε, την Αφρική, μια μεγάλη ήπειρο που αλλάζει πολύ γιατί έχουμε την να μιλάμε για την Αφρική, λες και πρόκειται για μια ενιαία περιοχή, λες και η Ευρώπη είναι ενιαία, για παράδειγμα. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τι θέματα θα είναι στην ημερήσια διατάξη στη συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αφρικανικής Ένωσης, η Επιτροπή και της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνδεθούν στις 22 Απριλίου να σας ενημερώσω για να συζητήσουν ακριβώς τα θέματα αυτά. Το Συμβούλιο έχει εγκρινεί συμπεράσματα για την Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται για τα θέματα αυτά και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο. 20 λεπτά. Και μετά θα ακούσουμε τους συναδέλφους για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ Λίντα. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που έρχομαι να σας μιλήσω. Δεν πρόκειται να σας ε, ταλαιπωρήσω και να μακρηγορήσω, γιατί θέλω βασικά να ακούσω τι θέλετε να ξέρετε εσείς για την Αφρική. Καλό θα ήταν να σας δώσω ωστόσο μια επισκόπηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης και τα θέματα ανάπτυξης και πώς εντάσσονται στο πλαίσιο των σχέσεων παντού ουσιαστικά με πάσα ειλικρινία. Οι σχέσει ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική ε, χρησιμοποιούν δύο ε, εργαλεία. Η Συμφωνία Συνθήκη του Κοτονού που καλύπτει οικονομικέ και πολιτικέ σχέσει μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του μεγαλύτερου δηλαδή τη πλειονότητα των χωρών τη Αφρική και ύστερα από την κοινή ε, στρατηγική Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης Jazz, όπως α, α, ονομάζεται. Το 2007 συνήφθη μεταξύ των Αφρικανικών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λισαβόνα. Η στρατηγική αυτή λοιπόν, η στρατηγική αυτή αποτελεί ένα πολύ συναπτικό έγγραφο που καλύπτει οκτω τομείς ε, επί παντός ε, του. Τον Απρίλιο πέρσι στις Βρυξέλλες, περίπου ένα χρόνο πριν, έλαβε χώρα μια σύνοδος Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεγαλύτερη που έχει λάβει ποτέ χώρα. Και έτσι ξανακοιτάξαμε όλη τη γκάμα της κοινή στρατηγικής αυτής. Και κοιτάξαμε πιο άμεσα τρία βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο υπήρων. Η ειρήνη, η ευημερία και η λαή. Αυτό ήταν επιβεβαιώθηκε στα συμπεράσματα της Συνόδου. Και θα κοιτάξουμε λοιπόν τι συμφωνήσαμε και τι κάνουμε τώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία αυτή των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής είναι, όπως είπε και η Πρόεδρος, η, η συναντήσει μεταξύ τη Επιτροπή τη Αφρικανική Ένωση και τη ε, Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. που θα λάβει χώρα στι 22 Απριλίου εδώ στι Βρυξέλλε. 9 από του 10 Επιτρόπου τη Αφρικανική Ένωση θα παρευρεθούν και 21 από του 28 Αντιπροέδρου και επιτρόπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επίση θα συμμετέχουν. Μεγάλη προσέλευση και αυτό καταδεικνύει τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ε, περιστασής. Η ε, κυρία Τζούμερ θα προετρέψει από πλευρά της Αφρικανικής Ένωσης και θα καλύψει σχεδόν το πλήρες ε, εύρος των σχέσεων μας θέματα ανάπτυξης, ειρήνης, ανάπτυξης, επιστήμη, γεωργία, έρευνα, εμπόριο, υποδομές, βιομηχανία. Θα υπάρχουν λοιπόν υποομάδες που θα καλύψουν σχεδόν όλα αυτά τα θέματα και όπως σας είπα θα τονίσω κάποια που θα έχουν προεξέχουσα σημασία. Σε κάποια φάση φέτος επίσης θα υπάρξει ένα κοινό ετήσιο φόρουμ σε επίσημο επίπεδο. Μία συνάντηση αποτελεί αυτή η περίσταση για να ελέγξουμε την εφαρμογή των συμφωνιών των ε, συνόδων. Κάποια στιγμή, κατά πάσα πιθανότητα, στις αρχές του φθινοπόρου στην Αμπέμπα και θα συμμετάσχουν και τα 54 κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης και 28 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δύο επιτροπές. Μεγάλη λοιπόν εκδήλωση η κοινωνία των πολιτών, η βιομηχανία, η οικονομία θα εκπροσωπηθούν προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα συμπεριληφθεί όλη η γκάμα των σχέσεων μεταξύ των δύο υπήρων. Η επόμενη σύνοδος μεταξύ των δύο υπήρων θα γίνει το 2017, τρία χρόνια μετά την τελευταία. Κάπου στην Αφρική. Δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς πού. Το δυνατό σημείο των σχέσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στα κοινά συμφέροντα αλλά και στις κοινέ αξίες και στους κοινούς στόχους. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν με αντίστροφη σειρά ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες. Οι σχέσεις λοιπόν έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μεταξύ των λαών. Αυτό εμπεριέχει διάφορες συνιστώσεις. Οι λαοί και οι επαφές, οι ενταλλαγές μεταξύ των λαών. Αυτό εμπεριέχει το όλο ζήτημα της μετανάστευσης. Θα επεκταθώ λίγο πιο μετά από αυτού. Κατά δεύτερον, την ανθρώπινη ε, ανάπτυξη, εκπαίδευση, υγεία, τέτοια θέματα τα οποία, που είναι απαραίτητα για την ε, εξέλιξη των ατόμων. Και τρίτον, τα δικαιώματα των ατόμων, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα μειονοτήτων, δικαιώματα, δικαιώμα έκφρασης, ε, συνεταιρίζεσθε, βασικές αξίες όπου υπάρχει πολύ πιο μεγάλη συμφωνία και κοινό τόπος από ό,τι μπορεί να αντιλαμβανόμαστε, γιατί τίνουμε να προβάλλουμε μόνο τα σημεία όπου δεν υπάρχει απαραίτητα συμφωνία. Για να επανέλθω στα θέματα της μετανάστευσης. Η μετανάστευση, η μετανάστευση αποτελεί ένα πολύ ένεργο θέμα και για τις δύο πλευρές και μία πρόσφατη διακήρυξη που περιλαμβάνει ένα πενταπλό σχέδιο δράση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρικανική ε, Υπήρου αναγνωρίζεται μετανάστευση ω ένα κοινό ζήτημα όπου και οι δύο Ήπειροι έχουν παρόμοια συμφέροντα. Ποια είναι λοιπόν τα παρόμοια συμφέροντα αυτά. Καμία από τις δύο Ήπειρους καταρχάς δεν θέλει να εξαναγκαστεί ο κόσμος να εξαναγκάζεται να μετακινείται λόγω πολιτικών ή οικονομικών συνθήκων. Όλοι θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά εκεί που επιλέγουν. Θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα μετακίνησης αν υπάρχουν λόγοι. Να μην υπάρχουν τεχνητά εμπόδια, αλλά δεν θα πρέπει να εξαναγκάζεται ο κόσμος να μετακινείται, να μεταναστεύει παρά τη θέλησή του. Και εδώ λοιπόν έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα. Υπάρχουν τεράστιες μεταναστευτικές ροές στην Αφρική. Εμείς ε, γενικά έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε στη μετανάσταση μεταξύ των υπήρων, αλλά υπάρχει και στο εσωτερικό της Αφρικής, της υπήρου, μεγάλη ροή μεταναστευτική. Συχνά έχουμε πολλούς ε, εκτοπισμένου καταναγκαστικέ ε, μετακινήσεις του πληθυσμού και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τη διαχείριση των ροών αυτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να υπάρξει σωστή συνεννόηση με τι χώρε προέλευση των με τις χώρες των μεταναστών, με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε δύο διαδικασίες. Τη διαδικασία Ραμπάτ για την ε, Δυτική Αφρική και για το κέρας και για την Ανατολική Αφρική την διαδικασία του χαρτούμ. Αυτό λοιπόν καλύπτει σχεδόν όλες τις σχέσεις με την Αφρική. Η διαδικασία του Ραμπάτ έχει ξεκινήσει πριν από 10-15 χρόνια και σημειώνει καλή πρόοδο. Πραγματικά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι λειτουργούν πολλές από τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας και η, η διαδικασία του χαρτόμ ξεκινάει την ίδια διαδικασία τώρα στο κέρας της Αφρικής. Αν δεν είχαμε σχέσεις με τις χώρες προέλευσης, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την αιτία, την πηγή του προβλήματος. Και σας είπα και επαναλαμβάνω ότι έχουμε την ίδια αντίληψη. Δεν θα πρέπει να εξαναγκάσετε ο κόσμος να φεύγει. Ο διάλογος λοιπόν περιέχει όλα τα ζητήματα που άπτονται τη μετανάστευση, με όλες ε, τις χώρες, ακόμα και τις χώρες που ο κόσμος εξαναγκάζεται να φύγει. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταπολεμήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις ε, αιτίες της μετανάστευσης. Προφανώς αυτό δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνο την ε, Υπηρεσία εξωτερική δράση, αλλά όλα τα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα στη Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων, DG Home. Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία και <coughs> μεταξύ του Επιτρόπου Αβραμόπουλου και της ε, κυρίας Μογκερίνη υπήρξε μια συνάντηση τον περασμένο Νοέμβριο Και τώρα να περάσουμε στα θέματα ευημερία. Το δεύτερο μεγάλο τομέα των σχέσεών μας που αποτελεί και τον πιο άμεσο τομέα ανησυχίας της Επιτροπής σας. Όπως σας είπα, ορίζεται από την συνθήκη του Κοτονού και εδώ η υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχει να δραματίσει σημαντικό ρόλο μαζί με τους συναδέλφους από την DG DEFCO που ε, ευθύνονται και έχουν αρμοδιότητα για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι όπου έχει αρμοδιότητα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, γιατί σύμφωνα με την συνθήκη σε κάποιους τομείς έχουμε συναρμοδιότητα με την DG προκειμένου να υπάρχει συνοχή σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές. Να ληφθούν υπόψη και η πολιτική και η οικονομική διάσταση, ε, αλλά και τα θέματα ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν αντιπροσωπείες στις χώρες αυτές και με τις ε, κυβερνήσεις των χώρων αυτών συνεργαζόμαστε, αλλά και με τους ε, εκπροσώπους της, των τοπικών κοινωνιών. Δεύτερον, ένα απόσπαστο τμήμα της συνθήκης του Κοτονού είναι μια σχέση η οποία βασίζεται σε δύο πόδια, αν θέλετε. Το οικονομικό, οικονομική συνεργασία και το πολιτικό που είναι ο πολιτικός διάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 8. Χωρίς τα δύο πόδια δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν θα περπατήσει αυτή η σχέση, τουλάχιστον όχι ε, όσο γρήγορα θα μπορούσε. Και αυτό είναι ένα στο κομμάτι των σχέσεων μας με όλες τις χώρες της Αφρικής, αλλά και των άλλων χώρων ΑΚΕ. Πολύ σημαντικός λοιπόν και ο πολιτικός διάλογος, διότι σε κάποιους τομείς παρέχουμε βοήθεια που εξαρτάται από την ε, καλή ε, διακυβέρνηση της χώρας από τον εταίρο μας, ιδίως ε, στον τομέα της δημοσιονομικής στήριξης, που είναι αποτελεσματική μορφή βοήθειας. Πρέπει όμως να βασίζεται στο ότι τα χρήματα αυτά <clears throat> θα πάνε για το στόχο που προβλέπονταν. Και έτσι θα δημιουργηθούν οι υποδομές και οι δυνατότητες για την ίδια τη χώρα. Απαιτείται γι' αυτό όμως και συνεπής πολιτική, μακροοικονομική προσέγγιση, αλλά και μικροεφαρμογή. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Υπάρχουν προκλήσεις ενίοτε και είναι απόλυτα σωστό ότι εσείς η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ, η Επιτροπή Ελεκτρικού προπολογισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο φυσικά και θέλουν να είναι βέβαιοι ότι όταν δίνουμε δημοσιονομική στήριξη τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τον προβλεπόμενο σκοπό. Ο πολιτικός διάλογος λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το ίδιο και ο έλεγχος ε, και οι διαδικασίες λογοδοσίας ε, και λογιστικού ελέγχου. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου μια χώρα, εταίρος, παρεκκλίνει από τις απαιτήσεις όπως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε για τη της δημοσιονομικής στήριξης, την οποία και λοιπόν παρακρατούμε. Με τον πολιτικό διάλογο λοιπόν μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στη χώρα για να επανέλθει στη σωστή τροχιά. Συγκεκριμένα δύο είναι οι χώρες, η Ουγγάντα, Εκεί είχαμε απάτη σημαντική ε, στη χρήση ε, κάποιων κονδυλίων από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δεν πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια προερχόμενα από άλλου ε, χρηματοδότες ήταν, αλλά και εμείς και οι άλλοι χρηματοδότε ε, αναστήλαμε τη δημοσιονομική στήριξη μέχρι να εντοπιστεί η πηγή τη ε, απάτης αυτής και να αναλυφθεί δράση για την αντιμετώπιση και τη συγκεκριμένη περίπτωση απάτης αλλά και με την λήψη μέτρων για να μην ξαναυπάρξει κάτι αντίστοιχο. Και μετά συνέχισε πάλι η δημοσιονομική στήριξη. Είχαμε λοιπόν μια ένα πολιτικό μοχλό μέσω του πολιτικού διαλόγου. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αν απλά δίναμε βοήθεια προγραμματική. Δεύτερη χώρα το Μαλάουι. Cashgate ε, ήταν αυτή η υπόθεση, όταν ε, ολοκλήρωσε τα καθηκοντά της κυρία Πάντες πριν από δύο χρόνια και εμείς και άλλοι χρηματοδότες αναστήλαμε την παροχή βοήθειας μέχρι να ε, γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις, να ληφθούν μέτρα και πρόσφατα, λιγότερο δραστικά θέλετε, είχαμε αναστείλει τη δημοσιονομική μας υποστήριξη προς την Κάνα, γιατί τα μακροοικονομικά κριτήρια δεν τα τηρούσαν. Εκεί είχαν δε, κάποιε κάποιες ε, ενδείξεις για απάτη, ε, κάποιοι ισχυρισμοί και έπρεπε όλα αυτά να ερευνηθούν. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου αναστολής ήρθαμε σε επαφή και με το Εθνικό Ταμείο και εφαρμόστηκε έτσι ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Νομίζω σε δύο-τρει μέρε θα συζητηθεί στο Προεδρείο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που θα βοηθήσει την κυβέρνηση τη Γκάνα, την ε, δημοσιονομική τη θέση και την οικονομική τη κατάσταση να αντιβελτιώσει, να βάλει τα πράγματα πάλι στη σωστή τροχιά. Αλλιώ δεν πρόκειται να εκταμιευθούν κονδύλια για να πάνε σε κάποια εργάτες φαντάσματα που δουλεύουν στο κρατικό τομέα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σχέδιο του πολιτικού διαλόγου και η ΑΕΔ μπορεί να διδραματίσει έναν βοηθητικό ε, χρόνο, χρήσιμο θα έλεγα, στο πλευρό της ΔΕΦΚΟ που έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή. Παρομοίω, βέβαια η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο του προγράμματό μα σε μια σειρά από αφρικανικές ε, χώρες είναι τα περί διακυβέρνησης. Εκεί παρέχουμε σημαντική στήριξη για την ε, δημιουργία θεσμών που θα παρέχουν ε, μια υγιή, μια στέρεη βάση και για την οικοδόμηση της δημοκρατίας αλλά και για τη δημιουργία ε, διακυβέρνησης αποτελεσματικής στον τομέα της δημοσιονομικής διαχείρισης, της δικαιοσύνης, ε, δημοκρατικών θεσμών, βοήθεια στις εκλογικές επιτροπές, κοινοβούλια και ό,τι άλλο ποθεί καρδιά σας. Αυτή είναι μια πολιτική δέσμευση και βέβαια έχουμε και το σκέλος της πρακτικής εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων για να είναι επιτυχημένα. Θα επανέλθω στις εκλογές στο τέλος. Μιλάμε για ευημερία και όχι για βιώσιμη ανάπτυξη. Για ποιο λόγο. Διότι σε αυτό το, σε αυτή, σε αυτό το κεφάλαιο, αν θέλετε, ε, δημιουργούμε και σχέσεις και επαφές και με τον ιδιωτικό τομέα και με τους ε, εμπορικούς παράγοντες, διότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής σίγουρα αποτελεί σημαντικό κομμάτι των σχέσεών μας. Νομίζω 250 δις ευρώ το χρόνο από τη μία και προς τη και προς την άλλη κατεύθυνση είναι ε, ο όγκος των συναλλαγών, των εμπορικών, τεράστια επένδυση όπως καταλαβαίνετε. Το σημαίνει ότι Ευρώπη και Αφρική είναι οι σημαντικότεροι, μεγαλύτεροι εταίροι. Κάποιοι άλλοι βέβαια πλησιάζουν κάποιες αναδυόμενες οικονομίες, αλλά προς το παρόν παραμένει σημαντική η σχέση αυτή. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της είναι ε, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές από την Αφρική. Γύρω στο 40% πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα ή προϊόντα προσθέμενης αξίας και όχι πρώτες ύλε. Αν δείτε τις ε, εισαγωγές της Κίνας, για παράδειγμα, την Αφρική είναι ε, κατά αποκλειστικότητα πρώτες ύλε. Εμείς όμως εισάγουμε προϊόντα προσθέμενης αξίας βοηθάμε την ανάπτυξη, ε, τη στηρίζουμε το μεταπητικό κλάδο, δημιουργούμε θέσει εργασία και σε άλλου τομεί, όχι μόνο στην εξορρυκτική βιομηχανία. Και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε και ε, αν δει κανεί μόνο του αριθμού, ε, τι σχέσει αυτή μεταξύ Ένωση και Αφρική μπορεί να το παραβλέψει το στοιχείο. Αυτά λοιπόν ε, για το σημαντικό αυτό κομμάτι των σχέσεών μας. Η τώρα και η ΔΕΦΚΟ συμμετέχουν σε δράσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Ε, όχι για τους εξωτερικούς μόνο, αλλά και για τους εγχώριους επενδυτές. Και δύο τις βασικές φράσεις ε, στο τελευταίο, στην τελευταία σύνοδο κορυφής ΕΕ Αφρικής ήταν ε, να περάσουμε από τη βοήθεια στις επενδύσεις ε, όπως έγινε μετατόπιση στην Ασία τον τελευταίο καιρό και δεύτερον θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε, να απελευθερώσουμε το επιχειρηματικό δυναμικό εντός Αφρικής. Αυτά λοιπόν είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία και της πολιτικής μας. Και φυσικά γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με τη ΓΔ Εμπόριο πολύ στενά και ελπίζω όλο και περισσότερο με τη ΓΔ Επιχειρήσεις, όπου ε, το δυναμικό είναι σημαντικό για την ε, βελτίωση των σχέσεών μας στον τομέα αυτό. Τελευταία πτυχή πάντα στο πλαίσιο τη ευημερία που ανέφερα, είναι η πρόθεση τη περιφερειακή ολοκλήρωση. Από δική μα εμπειρία στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι οι ολοκληρωμένε αγορέ μπορούν να επιταχύνουν και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη. Πολλέ αφρικανικέ χώρε δεν έχουν αγορέ κρίσιμη μάζα επαρκού ώστε να μπορούν να ε, αναπτύξουν ε, επιχειρήσεις μεταπητικές, έντασης εργασίας, άρα ακόμα πιο σημαντικό από ό,τι για την Ευρώπη, είναι απαραίτητο εκεί να δημιουργηθούν αγορές που θα είναι μία βάση για την βιομηχανική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των μέτρων Και έρχομαι τώρα στον τελευταίο τομέα τη εταιρική σχέση που είναι η ειρήνη. Εδώ η έμφαση είναι όλο και μεγαλύτερη. Γιατί έχουμε καταλάβει πόσο σχέση υπάρχει μεταξύ ε, της ε, ειρήνης και της ασφάλειας, της ανάπτυξης της ασφάλειας. Γιατί με την πρόληψη των συγκρούσεων, όταν ξεσπάνε κάποια συγκρούσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι αναπτυξιακέ μα προσπάθειε εν γέννη. Και αυτό μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου. Διαχείριση κρίσεων όταν ξεσπούν. Εκεί συνεργαζόμαστε πολύ στενά Χρησιμοποιούμε τον αναπτυξιακό μας περιπολογισμό για να βοηθήσουμε τους Αφρικανούς ε, να αναπτύξουν ε, τη δυνατότητα διαχείρισης της κρίσης από μόνοι τους. Ε, διπλωματικά, πολιτικά, είναι ενεργοί, πάρα πολύ δραστήριοι, ιδίω περιφερειακές οικονομικές κοινότητες και Αφρικανική Ένωση προσπαθούν και να επιλύσουν και να προλάβουν συγκρούσεις. Όμως από ηλικής πλευράς μέσω Τη διευκόλυνση για την ειρήνη, την Αφρικανική διευκόλυνση για την ειρήνη, African Peace Facility, η Ευρώπη παρέχει βοήθεια εκεί που απαιτείται λόγω της κρίσης κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί παραδοσιακά να προσφέρει ο ΙΕ με τις ενευτικές δυνάμεις, άρα σύγκριση, επίλυση συγκρούσεων, δυνάμεις επίλυσης συγκρούσεων. Άμσο στη Σομάλια είναι το μεγαλύτερο ε, παράδειγμα εν μέρει χρηματοδοτείται από το African Peace Facility και παρέχεται μέσω της Αφρικανικής Ένωσης, αλλά και στο Μαλί και αλλού έχουμε χρηματοδοτήσει ε, κάποιες αποστολές και στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Και προσπαθούμε και στο Τσάντ, στη Λίμνη εκεί, να καταπολεμήσουμε την Πόκο Χαράμ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος διχρηματοδότης που μπορεί να παράσχει τέτοια βοήθεια. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η επένδυση για την αρχιτεκτονική της ειρήνης και της ασφάλειας όπως τη λέμε, για να μπορούν και οι Αφρικανοί να επιλύουν τις συγκρούσεις με ταχύτερο τρόπο. Θα μπορούσα με τα χαρά να επισέλθω σε μεγαλύτερε λεπτομέρειε, αν αυτό σα ενδιαφέρει, και να επεκταθώ σε κάποιε περιφερειακέ συγκρούσει ε, όπου έχει παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα απόσπαστο κομμάτι τη παροχή χρήσεων στι ε, ε, μεγάλε λίμνε, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρέχουμε υποστήριξη από ανθρωπιστική αναπτυξιακή πλέον. Έχουμε την περιοχή του Σαχέλ επίσης, όπου έχουμε τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για το Σαχέλ και νομίζω ότι εκεί ε, ήταν τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής της ολοκληρωμένης της συνολικής προσέγγισης. Επενδύσαμε σημαντικά στην ανάπτυξη των οικολογικά και οικονομικά ευάλωτων και εύθραυστων περιοχών του Σαχέλ και της Σαχάρας, ώστε η τρομοκράτες ε, και ε, οι εγκληματικές ομάδες να μην είναι οι μόνοι που θα ασκούν δραστηριότητες εκεί. Και η Δημοκρατία επίσης έχουμε ένα trust fund του Μπακού, το ίδρυσε η ΔΕΦΚΟ σε συνεργασία με Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Και εκεί εργαζόμαστε μαζί με την αποστολή της ΚΕΠΑ ε, UMAM, UFOR, ε, όλοι αυτοί συνεργάζονται και με τη Μινούσμα στο ΙΕ για την ε, ειρήνευση, την σταθεροποίηση και μετά βέβαια θα παράσουμε και αναπτυξική βοήθεια. Τέλος, η Νιγηρία, μεγάλη πρόκληση για τις χώρες γύρω από τη λίμνη του Τσάντ είναι η Μπόκο Χαράμ. Το αποτέλεσμα των εκλογών ελπίζω θα οδηγήσει σε ανανεωμένη έμφαση στη προσπάθεια επιτάχυνση των οικονομικών εξέλιξεων στη Βόρεια Νιγηρία και ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, διότι χωρίς εκπαίδευση βλέπουμε πόσο μπορεί η Μπόκο Χαράμ να ε, διασπείρει το μήνυμά τη, να στρατολογήσει κόσμο και τελικά να πάρει στην κατοχή της και δάφη. Πρέπει λοιπόν να ε, προσθέσουμε και την κυβερνητική κρατική ανταπόκριση και την εκπαίδευση. Πάνω σε όλα αυτά Υπάρχει και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει την Επιτροπή Ανάπτυξη. Η πάροχη αναπτυξιακή βοήθεια ε, σε τέτοιου είδου έφραστε ε, συνθήκε σίγουρα συνεπάγεται κινδύνου. Πρέπει κανεί να πάρει ε, και κάποιο ρίσκο. Ότι μπορεί δηλαδή να χαθούν κάποιοι, κάποια χρήματα στην πορεία. βέβαια πρέπει να είναι ένα υπολογισμένο κίνδυνο, ένα πολιτισμένο ρίσκο αυτό. Και σίγουρα θα πρέπει να μπορούμε να παράσχουμε τα στοιχεία ε, που θα απαιτούνται. Αλλά αν δεν το πάρουμε αυτό το ρίσκο και η ανθρωπιστική βοήθεια θα ε, κατασπαταλάται και οι κρίσει θα επιδεινώνονται. Πρέπει να πάρουμε ένα ρίσκο για να σταθεροποιήσουμε μια περιοχή μετά από μια σύγκρουση. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο. Ποιος είναι ο στόχος μας. Να δημιουργήσουμε θεσμούς, διακυβέρνηση, για να μην ξαναπροκύψουν τέτοιες συγκρούσεις. Και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι και της αναπτυξιακής πολιτικής και της εταιρικής μας σχέσης με την Αφρική. Όπως είπα, έχουμε το κεφάλαιο διακυβέρνηση και επενδύουμε σε πολλούς θεσμούς, ε, ιδίως στις εκλογές. Είχαμε τις εκλογές στην Ιγυρία. Μόλις ε, επέστρεψα από εκεί, ήταν ένα κλασικό παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η Ιγυρία είναι μια τεράστια χώρα που μπορεί να τα καταφέρει, είναι αυτόνομη, να φτάξει, έχει πολλά χρήματα. Δεν θα σας πω τώρα πώς διανέμονται, δική τους ευθύνη είναι στη χώρα πώς το κάνουν αυτό, αλλά υπάρχουν παρόλα αυτά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και με την ε, πρόθεση των εκλογών παράσχομαι, παρήχαμε 35 εκατομμύρια ευρώ στην εκλογική επιτροπή, την ΑΝΕΚ και την κοινωνία των πολιτών τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, για την πρόθεση της εκπαίδευσης, της βελτίωσης των δυνατοτήτων, ε, τη δεξαγωγή των εκλογών, ε, παροχή εμπειριογνωμοσύνης. Monitoring. Πολιτική αγωγή, αγωγή του πολίτη και παρακολούθηση. επίσης, υπήρξε και επιτροπή, μάλλον αποστολή παρατήρηση εκλογών. Ο Σαντιάγο Φίσας ήταν ο επικεφαλής μαζί με μια ομάδα ευρωβουλευτών που ήταν εκεί ο Χαβιέρ Νάρτ ήταν ο επικεφαλής και ο ρόλος του ήταν άκρος απαραίτητος. Παρήχαν ανεξάρτητη αντικειμενική εξωτερική επαλήθευση. γιατί τη των εκλογών δεν ήταν μόνοι τους, Υπήρχαν αποστολές παρατήρησης από το ECOWAS, την Αφρικανική Ένωση, την Κοινοπολιτεία, USAID, NDI. Υπήρχαν και ντόπιοι παρατηρητές. Υπήρξε μια πολύ καλή προσπάθεια και συνεργασία Δηλαδή δεν αρκεί να έρθει ένας ε, και να πει τι καλή οι εκλογές και μετά μια άλλη ομάδα παρατηρητών να πει ε, χάλια πήγαν εκλογές. Ε, συνεργαστήκαμε πολύ καλά μαζί όλοι, συμφωνήσαμε τις συστάσεις και πραγματικά πήγε πολύ καλά η παρατήρηση των εκλογών και φάνηκε να πιστεύει ο κόσμος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είδαμε στην συνέντευξη τύπου. Τα προκατακτικά πορίσματα τα παρουσιάσαμε σε μια συνέντευξη τύπου που είχε τη μεγαλύτερη προσέλευση και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από, όλους, ε, από όλες τις άλλες παρατηρητών. Με όλες αυτές τις ε, συνδυασμένες μας δράσεις νομίζω ότι πραγματικά έχουμε συνεισφέρει στο να ε, ζήσει η Νιγηρία τις πιο δίκαιες και ελεύθερες εκλογές στην ιστορία της και είχαμε ιστορική αλλαγή, αλλαγή σκητάλη στην κυβέρνηση. Έχασε το κυβερνών κόμμα, κέρδισε το κόμμα της αντιπολίτευσης, έγινε η ε, αλλαγή αυτή με σχετική ειρήνη, θα έλεγα, ειρηνικά και ήρεμα. Ε, είναι πολύ ε, σημαντική αυτή η καμπή και νομίζω ότι και η στήριξη που μπορέσαμε να παρέχουμε και εμείς και πολλοί άλλοι βέβαια έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Και αυτό βοήθησε και την αποτροπή συγκρούσεων υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, πολύ πραγματικός ε, υπαρκτός κίνδυνος η μία πλευρά να προσπαθεί να κλέψει εκλογές ε, διαστρεβλώντας τη δικασία και αν γινόταν αυτό θα υπήρχαν εκατοντάδες νεκροί. Αυτό το αποφύγαμε και με αυτό, και με αυτό σταματώ και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με τα χαράς δε να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να υποβάλει ερωτήσεις για να ξέρω αν πρέπει να ανησυχώ για την ώρα. Um, Pedro Silva Pereira, Maria Heubuck, um, Mr. Weilenen, Heidi Hautala. So that's how many are? About yeah, seven, eight, six. Six. six. So about three minutes each. It's, it's... Γύρω στα τρία λεπτά έχετε έκαστος. Ο κύριος Βέντερ πρώτος. Βέντα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και εφόσον έχω μόνο τρία λεπτά να σας πω σύντομα εσείς περιγράψατε διάφορα στοιχεία ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής και των σχέσεων με την Αφρική. Αναφέρατε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά όπως η πολιτική σταθερότητα. Αναφέρατε ένα σωρό πυλώνες, εμπορικό, επιχειρηματικό, κοινωνία, ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικός διάλογος. Στο τέλος αναφέρατε την κυρία και θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στις ε, επερχόμενες εκλογές στο Μπουρούντι. διότι τελευταίως μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα στο, για, και το Μπουρούντι και οι επερχόμενες εκλογές δείχνουν ότι οι φόβοι των πολιτών είναι πραγματική. γιατί ε, δίνεται, ε, δίνονται διάφορε ερμηνείε στον εκλογικό νόμο. Οι διοργανωτέ των εκλογών λένε πω έχουν δίκιο, δίκιο και κάθε πολιτική, ε, πολιτικός αγώνας θεωρείται παράνομος. Επίσης η θέση της Εκκλησίας και η δραστηριότητα της Εκκλησίας δέχεται πειρά. Αυτά τα μηνύματα είναι σημαντικά και το στρατός αποκτά πολιτική σημασία. Άρα λοιπόν δημιουργούνται ένα σωρό ερωτηματικά για την κατάσταση στην χώρα αυτή. Οι επιπτώσει των όσων έγιναν στην Ιγυρία είναι πολύ θετικέ, αλλά το Μπουρούντι είναι μια από τις στοχότερες χώρες. Και γι' αυτό και η κατάσταση εκεί μπορεί να είναι πολύ διαφορετική και ανησυχητική. Το Μπουρούντι είναι πολύ σημαντική χώρα. Επίσης, τι ρόλο παίζουν οι πολιτικοί παρατηρητές των εκλογών, γιατί γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο πολιτικός διάλογος έχει να κάνει με την ε, πολιτική διαχείριση, κρατικά, τους κρατικούς θεσμούς και αυτοί οι θεσμοί αργά ή γρήγορα έρχονται και μας ζητούν αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι ο πολιτικός ε, αγώνας στη χώρα θα είναι ξεκάθαρος. Σας ευχαριστώ για την ε, εικόνα που μας δώσατε για τις σχέσεις της ε, Ένωσης με την Αφρική. Ίσως είναι μια λανθασμένη εντύπωση που έχω ότι όλα φαίνονται να είναι πολύ ρόδινα και αρμονικά με βάση ακούσαμε. Εγώ ωστόσο πιστεύω ότι πολλά έχουν να γίνουν, πρέπει να γίνουν στις σχέσεις ε, ένωσης με Αφρική. Υπάρχει έλλειψη σταθερότητας στην υποσαχάρη Αφρική, υπάρχει μεγάλη αποσταθεροποίηση στις χώρες εκεί και αποτελεί αυτό απειλή για τον κόσμο που ζει εκεί. Απειλές ε, από τη Δύση στην Ανατολή, Μαυρτανία, Κένια, Σομαλία, λείπει μια κοινή στρατηγική από πλευράς της Ένωσης ενώ εξαπλώνονται συγκρούσεις σε όλες αυτές τις περιοχές και που και που κάποιο μονομενο κράτος μέλος συμβάλλει λόγω ιστορικών δεσμών. Πάντως κοινή στρατηγική δεν φαίνεται να υπάρχει. Το δεύτερο που αναφέρατε είναι οι, οικονομικές, ε, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Μιλήσατε για τις πρώτες ύλε, τους πόρους που έχει η Αφρική, ε, να γίνεται η κατεργασία τους εκεί παρά να μεταφέρονται οι πρώτες ύλε κατέργασης στις βιομηχανοποιημένες χώρες. Αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες όμως και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης όσον αφορά τις πρώτες ύλε ε, στις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕΤ αναφέρατε εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Οι σχέσεις ανάμεσα στην ε, ΑΚΕ και την Ένωση τελευταία, τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια έχουν παραμεληθεί και έχουν αποδυναμωθεί. Για, μέχρι το 2020 θα πρέπει να προσβλέψουμε στο μέλλον και να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που έχουμε για να δώσουμε νέα όθεση σε αυτές τις σχέσεις και να εστιάσουμε περισσότερο ε, έμφαση στις ε, σχέσεις μας με τις χώρες αυτές της Αφρικής και της ε, Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς συνεργαζόμαστε με άλλους δωρητές όπως η Κίνα ή η Βραζιλία για την παροχή βοήθειας Ξέρω ότι η προσέγγιση των χωρών αυτών είναι πολύ διαφορετική, αλλά και εκείνοι προσφέρουν βοήθεια. Οπότε ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις. Και τέλος, σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ίσως πρέπει να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Παύελ Βάιλερ και μετά η Μαρία Χόιμπρουκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική σας εισήγηση. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με εκεί που τελείωσε τις παρατηρήσεις του κύριου Σεμόζερ, δηλαδή την, ε, τον ρόλο των άλλων ε, παιχτών στην Αφρική, πώς αναπτύσσεται η συνεργασία με τις ΗΠΑ στην αναπτυξιακή βοήθεια, έχουμε τον ίδια πολιτική προσέγγιση σε σχέση με τα πολιτικά προβλήματα της Αφρικής. Ποιος είναι ο ρόλος της Κίνας. Αναφέρατε την Κίνα ως ένα, μια χώρα που αγοράζει αποκλειστικά πρώτες ύλες από την Αφρική. Ποιος είναι όμως ο ρόλος της Κίνας στον αναπτυξιακό τομέα. ποιο είναι ο πολιτικό τη ρόλος και ε, βέβαια ξεχάσαμε την Ινδία που είναι ένας τρίτος μεγάλος παίκτη Ο κύριο Μαζέρο ανέφερε την Βραζιλία που είναι και αυτή σημαντική. Έχουμε λοιπόν Κίνα, Ινδία, Ηνωμένε Πολιτείε Ποιος είναι ο ρόλος τους. Ευχαριστώ. Κύριε Χόιμπρουκ. Και μετά ο Πέντρο Περέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Αφρικανική Ένωση χρηματοδοτείται κατά 90% από χώρες δωρητές και κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε πόσο εντατική είναι η οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Εδώ όμως θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Νόησερ, ο οποίος και αυτός διαπιστώνει ότι δεν έχουμε μόνο εμπαρικές σχέσεις για μεταποιημένα προϊόντα, έχουμε και πολλές πρώτες ύλες ε, οι οποίες έρχονται προς την Ευρώπη. Και αυτό σίγουρα αποτελεί ένα έλλειμμα από πλευρά μα. Η Αφρικανική Ένωση στην Αντίσα Μπέμπα τον Γενάρη άφησε και ψήφισε μάλλον ε, ένα μεγάλο όραμα με την ε, ατζέντα που υπερψήφισε. Τα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης φαίνεται ότι δεν ακόμα, δεν εμπιστεύονται ακόμα την ίδια τους την Ένωση. Και αυτό θυμίζει την Ευρώπη γιατί επί σειρά ετών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε περιορισμένε αρμοδιότητε. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εμείς έχουμε προχωρήσει πιο πολύ. Θα ήθελα να μας πείτε πώς ε, εκτιμάτε αυτό το νέο όραμα της Αφρική. Γενικά είναι καλό να υπάρχει όραμα, αλλά μήπω είναι υπερβολικά υψηλή η φιλοδοξία της Αφρικής σε αυτή τη φάση. Ε, εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το όραμα αυτό. Πρόκειται για ένα όραμα που θα επηρεάσει ενδεχομένω και την δική μας εταιρική σχέση με την Αφρική. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και άλλα σχόλια. Και τι θα γίνει μετά το 2020 με τη συμφωνία τη συνθήκη του Κοτονού. Θα αλλάξει, θα αποκτήσει μια νέα μορφή. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Ευχαριστώ. Πέτρο. Και μετά η Χάιντι, η οποία θα ξανάλθει. Και μετά και εγώ θέλω να πάρω το λόγο. Ο Πέτρο και μετά η Χάιντι, λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, προσκεκλημένο μας για την εισήγηση που μας έκανε για το πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική και να θέσω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η εξή. Εμεί ε, σε λίγε εβδομάδε έχουμε την διάσκεψη κορυφής της Αντίσα Μπέμπα, όπου θα αποφασιστεί το πλαίσιο χρηματοδότησης των πολιτικών ανάπτυξης μετά από το 2015. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι θα ήταν ε, μια, ένα καλό νέο στην διάσκεψη της Αντισαμπέμπας ή ε, ποια είναι τα πολιτικά μηνύματα και αποφάσεις που αναμένεται από αυτή τη διάσκεψη ώστε να μπορέσει να βοηθήσει και να προωθήσει τις αναπτυξιακές πολιτικές για την Αφρικανική Ήπειρο. Δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, των μεταναστευτικών ροών γιατί είναι ένα σημαντικό τμήμα της εταιρικής μας σχέσης με την Αφρική. Όλοι γνωρίζουμε τα δράματα που ζουν στην, που, που, που εξελίσσονται στην περιοχή της Μεσογείου με την διακίνηση μεταναστών Για τις διάφορες τραγωδίες που έχουν συμβεί. Θέλω να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγους για να είναι ικανοποιημένη με την ατζέντα της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης αυτών των μεταναστευτικών ροών στην Μεσόγειο με τρόπο ώστε στο μέτωπο του δυνατού να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια που βρίσκονται στην πηγή, στη ρίζα αυτών των ε, μεταναστευτικών ροών. Τρίτη και τελευταία ερώτηση έχει να κάνει για τις σχέσεις με τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Γουινέα Μπισάου και θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδοτική στήριξη προς τη χώρα αυτή. Η Γουινέα Μπισάου είναι μια χώρα που έχει νέα πολιτική ηγεσία με τον νέο Πρωθυπουργό Ντομίνγκο Σιμό Εσπερέρα και αξίζει μια ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσει να γυρίσει τη σελίδα της πολιτικής αστάθειας που έβλαψε πολύ την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Όπως γνωρίζετε η Πορτογαλία ε, παρακολουθεί για ιστορικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς λόγους από πολύ κοντά τις εξελίξεις ε, στην Γουινέα Βισάου και θα ήθελα να γνωρίσω ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι ε, αυτής της οικονομικής εταιρική σχέσης με την Γουινέα ΒΙΣΑΟ που είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Χάουταλα και μετά θέλω να πάρει το λόγο και η Έλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Εγώ έχω να κάνω ερωτήσεις για την συνεργασία για την ανάπτυξη και τα σχετικά εργαλεία. Αναφέρατε τη δημοσιονομική υποστήριξη και ποια αποτελέσματα μπορεί να πετύχει η δημοσιονομική υποστήριξη. Συμφωνώ ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο αυτό. Και πρόσφατος έχουμε δει στην Τανζανία ότι υπήρξε μια κατάσταση κακοδιαχείριση επασταλιών που οδήγησαν, αν δεν κάνω λάθο. σε μια κατάσταση αναστολή των πληρωμών. Θα μπορούσατε να μα εξηγήσετε Ποιος ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά δεύτερον, οι χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους και δεν είναι σε θέση ενδεχομένως να διαχειριστούν με διαφανή τρόπο τους πόρους αυτούς. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε χώρες όπως η Τανζανία, η Μοζαμβίκη και άλλες όπου υπάρχει η προοπτική εξωτερικής ε, βοήθειας σε 5 έως 10 χρόνια, αν τα πράγματα πάνε καλά και υπό τον όρο ότι θα μπορέσουν να εντρήσουν ισχυρούς θεσμούς που θα διαχειριστούν τις νέες αυτές ευκαιρίες. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας αναπτύξετε λίγο παραπάνω ποιε είναι οι απόψεις σας. Μία τρίτη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς αποτελεί μέλος της διεθνούς ε, εταιρική σχέση σε ό,τι αφορά τα ευάλωτα κράτη. Ποια είναι λοιπόν η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση αυτή και πώς σκοπεύετε να βοηθήσετε ιδιαίτερα τα ευάλωτα αυτά κράτη για να φροντίσουν τους λαούς τους. Ευχαριστώ, Γέλη Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ρωτήσω εν συντομία πώς έχει η κατάσταση για τον διάλογο πολιτικής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 της Συμφωνία Κοτονού και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΔ. Η Πρόεδρος, δύο πράγματα θα ρωτήσω. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε στα πλαίσια τη κοινή ε, συνεδρία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τα θέματα μετανάστευση. Μιλήσαμε λοιπόν για το θέμα το, της εκτορικής από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από την Αφρική. Εσά, ποια είναι η άποψή σα, ποια είναι η άποψη τη Υπηρεσία Εκτορική δράση και ποια πιστεύετε ότι είναι η αντίληψη που επικρατεί στην Αφρική Κάποιοι το συνέκριναν με την Αυστραλία και τις σχέσεις με την παππού Νέα Γουινέα. Τέτοιου είδους σχέσεις αναζητούμε. Και τώρα να σας πάρω από το κέρας της Αφρικής της Ζιμπάμπουε, όπου είχαμε δύσκολες σχέσεις πρόσφατα και πριν από κάποιες εβδομάδες από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται απόπειρες επανα... επανάληψη των σχέσεων με την χώρα. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν δύο λόγια. Μιλάμε για το θέσμα με την κυβέρνηση, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ποιοι ήταν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων. Τέλος, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση για την Κίνα και την Αφρική. Είναι λοιπόν μεγάλη σφαίρα επιρροή η Αφρική. Ο πρόεδρο Ομπάμα επισκέφθηκε την Αφρική, η Κίνα προσπαθεί να ασκήσει επιρροή. Πώ γίνονται αντιληπτέ αυτέ οι απόπειρε στην Αφρική. Θεωρούν ότι προσπαθούμε να αναμειχθούμε στα εσωτερικά του. Πώ επηρεάζουν αυτά τη δική του ατζέντα. Σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Θα προσπαθήσω να τι απαντήσω όλες τουλάχιστον συντομία και να προσπαθήσω να ακολουθήσω και μία σειρά. Ε, ε, ρωτήσατε για τις εκλογές για τον Μπουρούντι. Αποτελεί αυτό μια μεγάλη ανησυχία για μας. Όχι μόνο το γεγονός ότι γίνονται εκλογές, αλλά η δυνατότητα ο πρόεδρος Κουρουντίζα να προσπαθήσει να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Υπάρχει αντίθετη πολιτική συμφωνία Ακόμα και αν ε, υπό τεχνική άποψη το Σύνταγμα θα το επέτρεπε. Αυτό όπως είπατε, περιορίζει, συρρυκνώνει το πολιτικό φάσμα, το πολιτικό χώρο, καταπιέζει τους πολιτικούς αντιπάλους ε, και όντως μας ανησυχεί. Στην παρούσα φάση είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να αποστείλουμε μία αποστολή παρατήρησης των εκλογών, αλλά πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο ελεύθερων εκλογών. Ιδάλλω δεν έχει νόημα να στείλουμε την αποστολή. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε με σαφήνεια και με άλλους ε, πολιτικούς παραγοντές ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι πολιτικές δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την τρίτη θητεία. Και ξέρουμε ότι κι άλλοι το θέτουν το θέμα αυτό. Όχι μόνο από τις άλλες υπήρους, αλλά και από την ίδια την Αφρική, από τις γειτονικέ χώρες του Μπουρούντι. Πολλοί λοιπόν εξημών ε, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει όμως διαρκώς να ε, εξετάζουμε την κατάσταση αυτή και θα πρέπει να διασφαλίζουμε να, ότι θα πρέπει να θέσουμε το καλό παράδειγμα εκεί. Είχαμε μια σειρά καλών παραδειγμάτων πρόσφατα στις εκλογές στην Ιγυρία, επίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, ο πρόεδρος Καμπίλα θεωρούμε ότι ενδεχομένως να είχε δελεαστεί και αυτός από μια τρίτη θητεία ή να ήθελε να αναβάλει τις ε, εκλογές. Τώρα λοιπόν αναγκάστηκε να επιταχθεί ότι θα γίνουν οι εκλογέ το 2016 όπω αρχικά είχε προγραμματιστεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημάδια πρόοδο σε κάποιε ε, χώρε, αλλά ναι, όντω μα ανησυχεί η κατάσταση στον Μπουρούντι. Ο κύριο Νόιζερ, ήσασταν πολύ θετικό. Ε, ε, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Υπάρχει το θέμα της σταθερότητας από την ακτή του Ατλαντικού, Μαυριτανία, <coughs> μέχρι τη Σομαλία. Και Υπάρχει όλο και μια μεγαλύτερη ανησυχία ότι συνδέονται αυτές οι περιοχές που μας ανησυχούν. Έχουμε μια στρατηγική για το Σαχέλ και για το κέρδο της Αφρικής. Αυτό έχει συμφωνηθεί με τα κράτη-μέλη και έχουν συμμετάσχει και τα κράτη-μέλη. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να την εφαρμόσουμε, για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι συνεκτική προσέγγιση μας και ότι εφαρμόζουμε όλα τα εργαλεία μας την πλευρά της ανάπτυξης, τη ασφάλειας, στο πολιτικό σκέλος. Αυτό ήταν άλλωστε και ο στόχος της στρατηγικής αυτής. Η στρατηγική του Σαχέλ αναθεωρήθηκε από το τελευταίο συνέδριο εξωτερικών υποθέσεων εγκρίναμε το σχέδιο δράση του Σαχέλ. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα κράτη-μέλη για να αποτρέψουν τη ρίζος, παθηκοποίηση για να υπάρξει κοινωνία των πολιτών, να υπάρξουν θέσει εργασία για τους νέους, κάποια βασικά στοιχεία. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε να έχουμε ένα ευρύ φάσμα. Πάντα μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Επίσης προσπαθούμε να συμφωνήσουμε με τα Ηνωμένα Έθνη, άλλο ένα μεγάλο φορέα και με την Αφρικανική Ένωση. Η εκμετάλλευση των πρωτομελών αποτελεί βασικό σημείο ανησυχία. Η έκθεση Κοφιανάν για το Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατέδειξε ότι χάσαν τα τελευταία 10 χρόνια 8 δισεκατομμύρια ε, δολάρια. Λίγο πολύ σε διάφορες ε, συμβάσεις Κάνουμε επίσης ό,τι μπορούμε για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Και για την ε, Κεντροαφρικανική Ένωση το κάνουμε ήδη με τη διαδικασία Κίμπερλι για τα διαμάδια. Γνωρίζετε λοιπόν ποια είναι τα θέματα αυτά. Και ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές λύσεις το να βρούμε την ε, πιο αποτελεσματική λύση είναι το ευκταίο. Επίσης, διάφοροι βουλευτές έθεσαν το θέμα του κοτονού και το τι θα γίνει μετά το 2020. Η απάντηση είναι ότι θέλουμε να πούμε τη δική σας άποψη για το θέμα αυτό. Η πλευρά των χρόνων θα πρέπει να εκπληρώσει τους όρους που στους οποίους είχε δεσμευτεί να εκπληρώσει και θα ακολουθήσει δημόσια συζήτηση. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω ποιες είναι οι προσωπικές μου σκέψεις, αλλά αυτές είναι μόνο προσωπικές μου απόψεις. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να εκπνεύσει και να σταματήσει. Θα ήταν μεγάλο κρίμα, θεωρώ. Να εστιαστούμε πιο πολύ στις μεμονωμένους ε, τομείς. Κατά πόσο θα πρέπει να διευρυνθεί το παιδί εφαρμογή, να περιοριστεί. Υπάρχουν πολλά και βασικά ζήματα. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία αξία στην Συμφωνία του Κοτονού ω εργαλείο πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία συμπεριλαμβανομένης και αυτή ε, τη σύνδεση με τον πολιτικό διάλογο, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ε, διαχωρισμός. Είναι σημαντικό λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό. Άρα, προσβλέπουμε στη συζήτηση αυτή. Και εσείς, ε, Λίντα, μας ρωτήσατε ποιες είναι οι σχέσεις μας με τις αναδυόμενες οικονομίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τομέα αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερω που οι αναδυόμενε οικονομίε ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ για την Αφρική. Η Αφρική είναι μια χώρα που χρειάζονται όλο και πιο πολλέ επενδύσει. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Υπάρχει ένα καταμερισμό των εργασιών. Οι υποδομέ, για παράδειγμα, χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την Παγκόσμια Τράπεζα, από την Αφρικανική Τράπεζα και από την Κίνα που δίνει κάποιον ειδών πιστώσεις και κάνει μεγάλες κατασκευές ε, οδικών δικτύων, σιδηροδρομικών δικτύων, λιμένων. Πολύ σημαντικός λοιπόν ο κλάδος αυτός. Το χρειάζεται αυτό η Αφρική για να συνδέσει τις αγορές της και να υπάρξει παντού ανάπτυξη η Βραζίλα, η Βραζιλία και η Ινδία είναι εξίσου σημαντικοί φορεί. Και υπάρχει άλλος ένας ε, τομέας, ο οποίος συχνά παραμελείται. Όσο αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα στην Αφρική, τόσο αυξάνεται και η πολιτική συμμετοχή και η αντίληψη του τι χρειάζεται για να είναι βιώσιμε οι επενδύσει. Ένα παράδειγμα μόνο να σα δώσω, το οποίο είναι στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν. Η Κίνα επένδυσε σημαντικά ποσά στην πετρελαιοβιομηχανία και ω εκ τούτου έχει σημαντικά συμφέροντα όχι μόνο να διατηρηθεί η βιομηχανία αλλά και να αποτραπεί οποιαδήποτε σύγκρουση και στι δύο χώρε προκειμένου να μην υπονομευτούν οι επενδύσει τη. Άρα συνεργαζόμαστε στενά με την Κίνα για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε την ε, σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν. Πρόκειται για μία από τις χώρες που υποστηρίζουν τις προσπάθειες στα πλαίσια Άρα, από κάποιες απόψεις προσεγγίζουν οι μεν του δε σε τέτοια ζητήματα το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι έχετε εταιρικέ σχέσεις και μερικοί εξημών μπορεί να συμμετέχετε Δυστυχώς, όπως είπατε, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έχει πολύ πιο περιορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με τις δικές σας. Είναι ασύμετρη λοιπόν η σχέση. Είναι καλό ωστόσο που υπάρχει. Αποτελεί ένα σημαντικό φόρουμ για ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και για την δημιουργία σχέσεων με τις αφρικανικές χώρες. Αυτό είναι απαραίτητο για τις μακροπρόθεσμες ε, προσδοκίες και φιλοδοξίες. Η κυρία Χόιμπρουκ μας μίλησε για το όραμα του για το 2035 και αυτό σχετίζεται. Και είναι πολύ φιλόδοξο το όραμα για μια ενιαία ζώνη ρευτέρου εμπορίου στην Αφρική και αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει ένα βασικό κινητήριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη. Φυσικά οι οραματιστές είναι οραματιστές γιατί ακριβώς είναι η μειονότητα. Άρα κάποιοι θα πρέπει να προκριθούν και κάποιοι λοιπόν θα πρέπει να έχουν τη φιλοδοξία του οράματος. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο απότερος σκοπός μας, ακόμα και αν ξέρουμε ότι αυτό θα προαπαιτήσει πολύ καιρό και πολλά βήματα μέχρι να το πετύχουμε. Κύριε Σίβα Περέρα, μας ζητήσατε να σας πούμε ποιο είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2015. Αυτό θα ήθελα να μας το απαντήσουν οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Εγώ να σα πω την αλήθεια, δεν έχω χρήματα. Ε, μόνο πολιτική κάνω και απόψεις εκφράζω σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Δεν έχω αρμοδιότητα. Είναι περίεργο που φέτο είναι αντίστροφα τα πράγματα. Φέτο λοιπόν θα αντιστρέψουμε την κατάσταση. Πρώτα συζητάμε τα σχέδια και μετά κοιτάμε τα λεφτά. Να δούμε τι θα είναι το αποτέλεσμα για το θέμα τη μετανάστευση. Το θέσατε και εσεί, Πρόεδρε. Ένα παράδειγμα όπου η διαδικασία του Ραμπάτ είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι η Μαυρετανία σε κάποια φάση έφευγαν εκατοντάδε άνθρωποι από την Μαυρτανία ω παράνομοι μετανάστε. Και τώρα λοιπόν αυτό έχει σταματήσει ακριβώ γιατί έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια εταιρική σχέση κινητικότητα. Έχουμε δώσει χρηματοδότηση για δημιουργία θέσεων απασχόληση. Και στην τελική ανάλυση ούτε η ήταν ικανοποιημένη που έφευγε τόσο κόσμο για κάποιες αφρικανικές χώρες θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Και ότι δεν ανησυχούν και οι ίδιες για την ε, μείωση της εκροής μεταναστών. Και στην Κάνα, για παράδειγμα, όπου υπήρχε μεγάλη εκροή το 2005-2010. Και αυτό λοιπόν έχει είναι λοιπόν απαραίτητο να συνεργαστούμε με τις χώρες προέλευσης για να υπάρξουν συστήματα που θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες. Στην Κάνα, για παράδειγμα, 3.000 δολάρια κάνει για να διασχίσει κανείς στην Σαχάρα. Αν με αυτά τα 3.000 δολάρια δημιουργούνταν μια μικρή επιχείρηση, θα μπορούσαν να στεθούν πολλέ μικρέ επιχειρήσει που θα αφαιρούσαν όλο τον κόσμο. Αλλά εξωτερική ανάθεση τη ευθύνη αυτή δεν θα ήθελα, θεωρούσα ότι, ήταν, ότι είναι απόλυτα σωστό τρόπο. Υπάρχουν διάφορε ομάδε μεταναστών και είναι σημαντικό να κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχουν κάποιοι που είναι βασικά οικονομικές μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες και να ζητούν ευκαιρίες. Κάποιοι εξαναγκάζονται να φύγουν λόγω της φτώχεια, κάποιοι άλλοι όχι, κάποιοι προσπαθούν να φύγουν από καταστάσεις προσωπικής δίωξης. Αυτά θα πρέπει να τα αποτρέψουμε και Επίσης, αφρικανικές χώρες που έχουν προσυπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για τους πρόσφυγες έχουν τις ίδιες ευθύνες όπως και Και επίσης να πούμε ότι πολύ πιο πολλοί πρόσφυγες φιλοξενούνται μέσα στην Αφρική και υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ, στο Τσάντ, στο Καμερούν, στην Αθιοπία. Και είναι μεγάλο το φορτίο που επιβαρύνει τις χώρες αυτές ό,τι αφορά τη διαχείριση των προσφύγων. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν τους μετανάστες και τις πρόσφυγες με όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται. Γιατί τη Γουινέα μπισάω. Κάναμε ένα μια μεγάλη συζήτηση στην διάσκεψη των δωρητών την περασμένη εβδομάδα και μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε 1,1 δις ευρώ για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Γουινέα Μπισάο υπό τη νέα κυβέρνηση. Πραγματικό επίτευγμα. Έχουμε κυβέρνηση, έχουν, θέλουν να επενδύσουν, έχουν σχέδιο για το πώς το κάνουν. Υπάρχει συμφωνία για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας, κάτι το οποίο αναβαλόταν για χρόνια και η διεθνής κοινότητα είναι πρόθυμη να βάλει χρήματα για να συνοδέψει αυτή τη είναι πολύ ενθαρρυντική η κατάσταση. Βέβαια είναι μακρύ ο δρόμο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό με 160 ε, εκατομμύρια συγγνώμη, για τη γεωργία, όχι μόνο για το Κάσιου, αλλά ε, και για γενικότερα για την παραγωγή, για την τομέα της υγείας που είναι πίσω ε, και τρίτον διακυβέρνηση ε, γιατί πρόκειται για μια κυβέρνηση που ζητά βοήθεια ώστε να ανασυγκροτηθεί η χώρα. Ε, στοχεύουμε λοιπόν τη βοήθειά μας και προσπαθούμε να με την, με μια μεγάλη ομάδα δωρητών, διεθνών δωρητών για να επιτευχθεί αυτό. Τώρα, ε, και έτσι έρχομαι να, στα όσα είπε η κυρία Χάουταλα. Πώς χρησιμοποιούμε τις αρχές ε, που ισχύουν για να βοηθήσουμε ένα άλλο μεταβατικό κράτος στη Σομαλία. Εμείς ηγηθήκαμε στο να συγκεντρώσουμε μια, και να συντάξουμε μια σύμβαση οικοδόμησης κράτους ε, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για να φτιαχτεί ένα κράτος από το μηδέν στην ουσία. θέλουμε να ενισχύσουμε βασικές υπηρεσίες, βασικούς θεσμούς όπως το δικαστικό σώμα. Επίσης συνεργαζόμαστε για την ασφάλεια στην αυσιπλοεία. Είναι ένα καλό παράδειγμα όπου οι αρχές μουσεών έχουν αρχίσει να λειτουργούν. Προσπαθούμε το ίδιο και στο Νότιο Σουδά, αλλά πρέπει να πω ότι δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Ίσως υπήρχαν μεγαλύτερες εντάσεις. Προσπαθούμε να κάπως να τα καταφέρουμε, να, να, να μπορέσουν οι κοινότητες να συμβιώσουν καταρχήν. Δεν λειτουργεί πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι αρχές μπορούσαν να είναι πολύτιμες ε, ε, για ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης ρωτήσατε για την οικονομική διαχείριση και πάλι οι συνάδελφοι Ντεύκο είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το πώς λειτουργούν όλα αυτά. Το Νότιο Σουδάν είναι ένα παράδειγμα που μέχρι ότου να έχουμε σωστή οικονομική διαχείριση δεν θα σταματήσει η σύγκρουση, γιατί η σύγκρουση αφορά την πρόσβαση στους ε, πόρους της πετρελοβιομηχανίας, δηλαδή σε χρήμα. Ο κόσμος αυτό θέλει, να, να βάλει το χέρι στο χρήμα και μέχρι του να έχουμε τρόπο να ελέγξουμε ε, την ε, χρήση αυτών των ε, αυτού του ρευστού υπέρ προς όφελος του κόσμου η σύγκρουση συνεχίζεται. Τώρα για την Τανζανία και εκεί όπως και αλλού έχουμε προσπαθήσει να συνεργαστούμε όσο γίνεται πιο στενά με τους άλλους βασικούς δωρητές ε, και ιδιαίτερα εκείνους που στηρίζουν τον προϋπολογισμό όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, κάποια ε, κράτη-μέλη διμερώς και γι' αυτό είναι πολύ αποτελεσματική η κατάσταση. Στην Τανζανία μαζί με την εγχώρια πίεση, όπου γιατί το Κοινοβούλιο παίζει κρίσιμο ρόλο στο να επιβάλλει τον πρόεδρο του ΣΑΚ και τους ε, υπουργούς, μπας πάση συνδυασμένε προσπάθειε ε, τελικά επηρεάζουν την κατάσταση. Το θέμα τώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινότητας των ΛΟΑΔ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολιτικού μας διαλόγου παντού. Δεν είναι ο διάλογος αποκλειστικά γι' αυτό, είναι, καλύπτονται ένα σωρό θέματα, χώρια και διεθνή και περιφερειακά, οικονομικά, πολιτικά, αλλά και ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι που διαρκώς θίγουμε. Ε, προσπαθούμε που μπορούμε να συνεργαστούμε με ομάδες εντός των χωρών που προσπαθούν να προστατεύσουν αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε δηλαδή να συνεργαζόμαστε με τους ε, ντόπιου. Ε, η θανατική ποινή είναι ένα καλό παράδειγμα. Σε πολλές από αυτές τις χώρες υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν ενώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ κτλ. που επίσης υποστηρίζουν ε, το εγκατάργηση του ανατικής ποινής και το στηρίζουμε. Τώρα αυτοί πρέπει να πείσουν τις κυβερνήσεις τους βέβαια. Τώρα για τους ΛΟΑΔ προσπαθούμε ρητά να συνδέσουμε τα δικαιώματα αυτής της κοινότητας με τα δικαιώματα του ατόμου. τα βασικά δικαιώματα στα οποία έχουν συνυπογράψει περισσότερε αφρικανικέ χώρε. Γι' αυτό και είναι ένα από τα πιο εμφισβητήσιμα θέματα, τα πιο επίμαχα θέματα. Ε, και τελικά φτάσαμε σε μια καλή διατύπωση στην, διάσκεψη, στην Αφρικανική Διάσκεψη Κορυφής για την προστασία των ε, μειονοτικών ομάδων και αυτό θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε για να υποστηρίζουμε την ε, εξάλληψη των διακρίσεων κατά αυτής της κοινότητας. Και τέλος, Ζιμπάμπουε. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία επανάληψης των συζητήσεων και των, των επαφών με την κυβέρνηση της Ζιμπάμπου τα τελευταία 5-6 χρόνια όπου σταδιακά ε, ήρθαν τα περιοριστικά μέτρα και πέρσι μάλιστα τον Νοέμβριο συμφωνήσαμε με τα κράτη-μέλη ότι θα καταργήσουν και οι περιορισμοί του άρθρου 56, πράγμα που μας διευκολύνει να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση για να προετοιμάσουμε το δαπάνηση των, του προγράμματος, του σχετικού προγράμματος, σημαίνει τον εντοπισμό των τομέων που πρέπει να στηριχθούν. Υπάρχει ένα τομέα όπου θέλουμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση και δύο τομεί όπου θέλουμε να συνεργαστούμε με διεθνείς οργανισμούς ή άλλους φορείς εκτός της κυβέρνησης. ένας τομέας όπου συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση είναι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Ε, ο δικαστικό τομέα είναι ένα ε, τομέα όπου στη Ζιμπάμπουε έχει αποδείξει ένα βαθμό ανεξαρτησία και θέλουμε αυτό να το ενισχύσουμε δίνοντας κάποια ε, στήριξη. Αλλά το βασικός όγκος των χρημάτων μας δίνεται στον τομέα της υγείας και εκεί συνεργαζόμαστε με τη UNICEF, άλλους ε, οργανισμούς, ε, ΜΚΟ κτλ. Οπότε τα χρήματα δεν περνάνε μέσα από την κυβέρνηση. Αν και είναι ένα τομέα που έχουμε συμφωνήσει με την κυβέρνηση ότι είναι προτεραιότητα. Και αυτό είναι τμήμα τη σταδιακή μα επαφή. Ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το λαό τη χώρα. Εκεί όπου μπορούμε το κάνουμε σε συμφωνία με την κυβέρνηση. Νομίζω πως έτσι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Α, ναι, είπα. Υπάρχουν δύο τομείς, ένας πολιτικός και ένας ασφάλειας. Η Άμισον στηρίζεται με τρεις τρόπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα επιδόματα στους ε, στρατιώτες, Ο ΙΕ την ε, υλικοτεχνική μέρημνα και η ΕΠΑ την κατάρτιση και το, το, βασικό υλικό ε, και ε, εκεί σιγά σιγά ε, μπορέσαμε να διώξουμε το Al-Shabaab. Στην Ιγυρία από που έρχομαι επίσης συνεργαζόμαστε με τη ΣΥΠΑ για να στηριχθεί το πρόγραμμα δράσης και συνεργαζόμαστε στενά για να δούμε πώς θα ε, καταπολεμήσουμε τον πόκο Χαράμ. Έχουμε πολλά που μπορούμε να κάνουμε στην ασφάλεια οι συνάδελφοι τη ΔΕΦΚΟ πούμε, μπορούν να σας πούν ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά στον τομέα τη υγεία ε, λόγω της δέσμευσή του και τη εμπλοκή τους στον τομέα του AIDS. Εμείς δεν δαπανούμε λοιπόν χρήματα εκεί, άρα γίνεται μια κατανομή εργασία. Εμεί ε, ε, εμείς βοηθάμε περισσότερο σε άλλους τομεί. Σε κάποιου τομεί λοιπόν συνεργαζόμαστε, σε άλλου μοιραζόμαστε τη δουλειά. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Σας, ε, να ευχαριστήσουμε τον ε, κύριο Ρίσκοτ για τον ε, μεγάλο αυτό περίπλου. Στην Αφρική πιθανότατα θα πρέπει να επανέλθουμε σε πιο συγκεκριμένα σημεία. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Αφού μόλις επιστρέψατε από την Νιγηρία, οπότε σίγουρα έχετε κερδίσει την ξεκούρασή σας στη διάρκεια των Πασχαλινών διακοπών. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Okay, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελευταία μέρα πριν ε, τις πασχαλινές διακοπές, αλλά μένουν δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο, πολύ σημαντική έκθεση, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή πριν την συνεδρίαση του Ιουλίου στην Αντισαμπέμπα. Λέμε τι θέλουμε να, ε, ποια θέλουμε να είναι η έκβαση αυτής της διάσκεψης. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Αν συλλέγονταν περισσότεροι πόροι θα διπλασιαζόταν ένας η αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Έλλη Σλάιν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας για τη φοροδιαφυγή και φορο για γιατί διακυβέρνηση ως προκλήσεις για διακυβέρνηση, κοινωνική προστασία και ανάπτυξη. Έχουμε την χρηματοδότηση ανάπτυξης βέβαια και τη σχετική διάσκεψη να τη ΑΜΠΕΠ. Συμπληρώνεται και η έκθεση του κυρίου Σίλβα Περέιρα. Πάρα πολύ σημαντική η διάσκεψη γιατί θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα αυτής της ε, διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και η έκβαση άλλων μελλοντικών. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε τα αποτελέσματα και τους επιδιωκόμενους στόχους. Έχουμε τους νέους στόχους για την ανάπτυξη. Η επίσημα ανάπτυξη και βοήθεια θα πρέπει να παραμείνει σημαντικό πυλώνας, να χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά. Δεν μιλήσουμε όμως μόνο για αυτό, αλλά και για την κινητοποίηση εθνικών πόρων που πρέπει να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Τα, ε, οι εγχώριοι πόροι θα συνεχίσουν να είναι το βασικό πόρο χρηματοδότηση για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Αλλά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή είναι τεράστιο εμπόδιο. Οι ροέ παράνομων κεφαλαίων είναι περίπου δεκαπλάσιοι των ροών βοήθειας που φτάνουν στις χώρες. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές, ε, σημαντικά φαινόμενα ε, ανάπτυξης, αλλά να επηρεάσει και τη διακυβέρνηση και τη δημοκρατικούς θεσμούς. Όμως υπάρχουν όρια στο τι μπορούν να επιτύχουν από μόνες τους οι χώρες, ιδιαίτερα για τις χώρες που δεν έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες όσον αφορά την ε, φορολογική ε, δομή και διαχείριση. Αφού έχουμε απαριθμίσει όλες τις δυσκολίες και τους οικονομικούς, πολιτικούς, διοικητικούς δεσμούς, που, ε, μάλλον ε, ε, φραγμούς που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροφυγής, θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ένα πρόγραμμα δράσης για να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή και να δημιουργήσουν πιο στέρεα και δίκαια φορολογικά συστήματα. Προσπάθησα να Τονίζω 10 βασικά σημεία και θέλω να συνεργαστώ με τους κοιόδες εισηγητές για να ε, μπορέσουμε να τα συμπληρώσουμε αυτά τα σημεία. Να σας αναφέρω κάποια σημεία που πιστεύω θα υπάρχει συνένεση. Καταρχήν η Κομισιόν θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες παρέχοντας τεχνική και οικονομική βοήθεια γιατί η βοήθεια, σε αυτούς τους τομείς είναι χαμηλή. Το 2011 ήταν λιγότερο από το 1% ολόκληρης της αναπτυξικής βοήθειας. Στον τομέα του πολιτικού διαλόγου θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στη ορθή διακυβέρνηση σε θεωρολογικά θέματα και να εγγυηθούμε ισότιμη κατανομή των δικαιωμάτων και τη φορολόγηση όταν μιλάμε για ε, συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Επειδή θα πρέπει να δοθεί το καλό παράδειγμα ορισμένων ε, ε, κρατών ε, και την επιρροή των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, στις αναπτυσσόμενες αυτές χώρες. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν πλήρεις και δημόσιες ε, πληροφορίες για την ownership ιδιαίτερα για να αποφευθούν οι επιχειρήσεις σε φαντάσματα όπου κρύβονται η φοροδιαφυγή ή η παράνομη χρηματοδότηση τρομοκρατίας, γενικά διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι ε, που σε αυτή τη κατάσταση είμαστε κάπως περιορισμένοι και ε, μπορεί να μην ε, ωφελήσει τελικά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ιδιαίτερα υπάρχουν δύο βασικά στη μέσα. Μιλάω για το country by country reporting και για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που θα έπρεπε να οικοδομηθούν λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις απαιτήσει των αναπτυσσόμενων χωρών. Στην ε, αναφορά αναχώρα πρόκειται για χώρες εκεί που λειτουργούν οι πολυεθνικές και που θα έπρεπε να έχουμε ε, εις βάθος πληροφορίες για να έχουμε μια αρχή σταθερή ότι δηλαδή οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργείται το κέρδος και θα πρέπει να προβλέπεται μια μεταβατική περίοδο για τις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν έχουν ε, πλήρως αναπτύξει τις υποδομές και τις απαραίτητες δυνατότητες για να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να μοιράζονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο είναι η δημιουργία ενό διακυβερνητικού οργανισμού για να εγγυηθούν ότι οι χώρε οι αναπτυσσόμενε θα συμμετέχουν ισότιμα στη μεταρρύθμιση του γενικού φορολογικού συστήματο. Για παράδειγμα, με την συμμετοχή της ειδική Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ. Και τέλος, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα θέματα του φύλου και όταν μιλάμε για φορολογική δικαιοσύνη. Γιατί τα χρήματα που λείπουν λόγω της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής είναι απαραίτητη πόρη για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι πολίτες της κάθε χώρας με προφανή επίδραση στα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας που είναι συνήθως οι γυναίκες. Άρα λοιπόν ε, θέλω να συνεργαστώ με τους σκιώδεις και είμαι βεβαία ότι το Κοινοβούλιο θα συντάξει μια ξεκάθαρη έκθεση με ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ώστε να επηρεάσει τη διαπραγματεύσεις στην Βέβαια και να δώσει κίνητρα και να παρατρύνει και την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you, thank you very much for that. Um, we have the shadow... Σας ευχαριστώ. Έχουμε σκιώδεις εισηγητές. Ρούμπιχ, πρώτος και έπονται άλλοι. Λιούκε, ναι. Τέλο πάντων, έχουμε. Τη Χάιντ επίση. Παύλο Ρούμπι, πρώτο. Ευχαριστώ. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Έλλη Σλάιν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στα σημεία εκεί όπου υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και γνωρίζουμε ότι 1,2 δις ανθρώπων ζουν με λιγότερο από ένα ευρώ τη μέρα. Θα σου πρέπει να τα βγάλουν πέρα. Και πάντοτε το ίδιο πράγμα χρειάζεται, ε, υποδομές, υγεία, παιδεία, και απασχόληση, ε, λογική αξιοπρεπής απασχόληση. Έχουμε αυτό το στόχο 0,7% του ΑΕΠ. Είναι ένα σημαντικός ε, βασικός στόχος, αλλά ακόμα πιο σημαντικό κατ' είναι να δούμε πώς ε, μπορούμε να συνδυάσουμε τους δημόσιους χώρους με τους ιδιωτικούς και νομίζω ότι ακριβώς αυτή η μικροχρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει και το blending, η ανάπτυξη δηλαδή θα μπορούσε επίσης να έχει μια πολύ πιο αποτελεσματική συνεισφορά στην καταπολέμηση της στόχιας. Εάν δούμε περίπου τι γίνεται το χρόνο, να 3 ευρώ ξέρουμε ε, πηγαίνει σε παρολογικούς παραδείσους ε, και σε εταιρείες ε, εξωχώριες πρέπει να συγκρίνουμε το ποσό αυτό με την αναπτυξιακή βοήθεια. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ώστε να μειώσουμε αυτό το χάσμα. Και επίσης ε, συμφωνώ απόλυτα με την ε, εισηγήτρια ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τους φόρους. Και τα κέρδη να παραμένουν ε, στην ε, Ένωση. Θέλουμε το ίδιο βέβαια να ισχύει και στις αναπτυσσόμενες. Υπάρχει και η τεχνική βοήθεια που είναι πολύ σημαντική, υπάρχει πολιτική γειτονία που ίσως θα μπορούσε να ε, κύπτει σε κάποιες πρωτοβουλίες αδελφοποίησης, κατάρτισης υπαλλήλων, παροχής επιτόπου εκπαίδευσης. Απόκτηση γνώσεων. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για τις ε, αφρικανικές και ασιατικές χώρες. Έχουμε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλες τις χώρες της ε, Αλλά υπάρχει το πρόβλημα της διαφθοράς και δεν φτάνουν τα χρήματα εκεί που έπρεπε να πηγαίνουμε Τι τις υπηρεσίε. υπηρεσίες όμως μπορούμε να έχουμε επαγγελματίες, ικανούς, ε, υπαλλήλου και στατιστικές υπηρεσίες που θα βλέπουν τι γίνεται ακριβώς. Και νομίζω ότι χάρη σε αυτού του είδους επενδύσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά και θα, να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα, την Κορέα. Στην ε, Βόρειο Κορέα ακόμα ο κόσμος πεινάει γιατί υπάρχει ένα δεκτορικό κομμουνιστικό σύστημα το οποίο αφήνει τον κόσμο να πεινάει και να πεθαίνει από την πείνα. Έχουμε στην Νότια Κορέα ένα δημοκρατικό σύστημα, ε, μια οικονομία της αγοράς ε, η οποία έχει καταστεί πλέον βιώσιμη και πλέον συνεισφέρει στην αναπτυξιακή πολιτική. Βλέπουμε λοιπόν τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ συστημάτων. Πιστεύω επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να προωθηθούν και θα πρέπει να είναι εξάρτητες. Έχουμε στην Ευρώπη το πρόγραμμα των Business Angel, των επιχειρηματικών αγγέλων. Θεωρώ ότι και αυτό αποτελεί προτεραιότητα και θα ήθελα να υποστηρίξω από την εισηγήτρια την κυρία Σλάιν. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί οι γυναίκε επιχειρηματικέ άγγελοι επίση θα πρέπει να τονιστούν. Πιστεύω ότι στην αναπτυξιακή πολιτική αυτό μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Και δυστυχώ ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνουμε πολλά υποστηρίξη. Η Επίτροπο ε, ε, καθυστερεί το πρόγραμμα αυτό και θα θέλαμε λοιπόν τα προγράμματα αυτά να προωθηθούν και στην Ευρώπη αλλά και στις αναπτυσσόμενε χώρε με την σχετική τεχνογνωσία βέβαια. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Ο κύριος Λούκη τώρα έχει το λόγο. Και η κυρία Χάουτολα στη συνέχεια. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τι εργασίε μα, η έκθεσή τη. Το θέμα είναι προφανές το πρόβλημα είναι προφανέ, Ε, υπάρχει μεγάλη συνένεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που έχει γράψει στην έκθεση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες πιο επιμέρους πτυχές όπου έχω διαφορετική άποψη. Αφενός φαίνεται ότι εξειδανικεύονται κάπως οι αναπτυσσόμενες χώρες σε ό,τι αφορά την παρουσίαση προβλημάτων. Παρουσιάζονται ως ε, καλά κράτη, καλές κυβερνήσεις, οι οποίες ε, δεν μπορούν να έχουν αρκετά φορολογικά έσοδα. Δίνεται η εντύπωση ότι τα φορολογικά έσοδα σχεδόν αυτονόητα χρηματοδοτούν υποδομές, ε, εκπαίδευση και άλλους ευγενείς σκοπούς. Είναι λίγο αφελές αυτό. Ίσως θα πρέπει να το διευκρινίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στις χώρες αυτές είναι ότι τα φορολογικά έσοδα εξυπηρετούν άλλους σκοπούς αυτές τις χώρες από αυτούς που θα θέλαμε στην έκθεση. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στην ε, αγοραστική δύναμη των ε, κρατών αυτών είναι ότι το προλογικό σύστημα είναι λάθος ε, από την αρχή και, και οι φορολογικές υπηρεσίες είναι λαπτωματικές και φυσικά υπάρχει και το θέμα της διαφθοράς όπως αναφέρθηκε στη δημόσια διοίκηση. Άρα δεν ε, συμφωνώ με την ε, εκτίμηση για την εμπορική απελευθέρωση όπως περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή και σε ό,τι αναφέρεται με τη μείωση των κρατικών εσόδων. Ξέρουμε ότι η τελωνιακή δασμή είναι ένας πολύ ελλειπής τρόπος για κρατικά έσοδα και δεν θα έπρεπε να τον υποστηρίξουμε. Ξέρουμε ότι η απελευθέρωση του εμπορίου έχει και θετικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα έσοδα του κράτους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επί της αρχής, δηλαδή, θα χρειαζόταν ε, μια αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος που θα καταργούσε τους δασμούς για το διασυνοριακό εμπόριο και θα κινούταν προς μια μοντέρνα διαμόρφωση, σύγχρονη διαμόρφωση της φορολόγησης των ε, χώριων προϊόντων. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να βάλω ένα ερωτηματικό εκεί όπου μιλάτε για την ε, στενή φορολογική βάση και λέτε ότι αν διευρυνθεί η φορολογική βάση θα είναι δυνατόν να έχει πιο πολλά έσοδα το κράτος. Θα ήθελα να επίσης την προσοχή σας στο εξή. Η μικρή φορολογική βάση στις αναπτυσσόμενες χώρες συνοδεύεται με εξαιρετικά υψηλό φορολογικό συντελεστή για τη μικρή αυτή βάση και αν διευρυνθεί η φορολογική βάση που είναι σωστό ο στόχος θα πρέπει να μειωθεί ο φορολογικός συντολευτής γιατί θα προκαλούνταν διαφορετικά μεγάλες στρεβλώσεις στο κάθε οικονομικό σύστημα και αυτό είναι φυσικά κάτι απευκταίο. Σε κάποιες περιπτώσεις η έκθεση αναφέρει ότι οι φόροι είναι πολύ πιο χαμηλοί στις αναπτυσσόμενες χώρες από τις και ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια εξίσωση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει δικαιολογημένο, δικαιολογημένα οι συγκεκριμένοι συντελεστές στις φορές. Και είναι μικρή φορολογία γιατί λίγα, λίγες είναι οι κοινόφελες υπηρεσίες που προσφέρονται. Η σχετική έκθεση που εγκρινάμε σε μηνύο μέλη την προηγούμενη εβδομάδα το επισήμωνε αυτό ρητά και θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και εδώ αυτή η ιδέα. Είναι φυσιολογικό το γεγονός ότι είναι πιο χαμηλό το φορολογικό φορτίο στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό δεν είναι κατά βάση κάτι ταπευκταίο γιατί χρησιμοποιούν λιγότερα το σύστημα το δημόσιο, έχουν μικρότερη ασφάλεια, κοινωνική ασφάλεια, υγειονομική ασφάλεια. Και αυτό συνοδεύεται με ένα χαμηλό επίπεδο φορολόγησης. Το ότι η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εκεί που γίνεται και δημιουργείται το κέρδος, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Η έκθεση εδώ προσπαθεί να κατακρίνει ατασταλίες, πασιφανείς ατασταλίες. Σύμφωνο. Αλλά ένα πρόβλημα της φοραποφυγής είναι το εξής. Η δημιουργία υπεραξίας στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες με διάφορα τεχνάσματα φορολογικά μεταφέρονται τα κέρδη σε φορολογικούς παραδείσους. Εκεί γίνεται μια εικονική φορολόγηση με πολύ χαμηλούς συντελεστές, χωρίς ουσιαστική δικαιολογία η ουσιαστική φορολόγηση στις χώρες αναπτυσσόμενες. Δύο άλλα ζητήματα. Η μελέτη αντικτύπου. Ποια είναι ποιες είναι οι συνέπειες στις υποανάπτυκτες χώρες. Θεωρώ ότι καλύτερα θα ήταν να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για να αυξήσουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες τις δυνατότητες φοροσυλλογής και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του της ε, συνθήκης προλόγησης του ΟΗΕ. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, δεδομένο ότι υπάρχει η ορμή σήμερα για το μοντέλο του ΑΟΣΑ. Και εφόσον ακολουθούμε το μοντέλο του ΟΣΑ, δεν έχει νόημα να ακολουθούμε παράλληλα δύο μοντέλα. Και καλά θα έκαναν οι αναπτυσσόμενε χώρε να ακολουθήσουν τα σφαίροντά του στα πλαίσια του ΩΣΑ. Ε, Κυρία Χάουταλ, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο σύντομη. Καταρχά, θα ήθελα να πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το σχέδιο έκδοση Έλλη είναι πολύ καλό δεν είμαστε αντίθετοι με κανένα από τα σημεία αυτού του σχεδίου έκθεση. Αντιθέτω θα θέλαμε να διευκρινίσουμε και να προσθέσουμε και κάποια καινούργια ε, στοιχεία. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για την αναφορά αναχώρα ω υποχρέωση των πολιοθνικών εταιριών, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί ότι η σημερινή υποχρέωση ε, του τραπεζικού τομέα θα πρέπει να επιταθεί σε όλους τους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο όταν μιλάμε για μια συνεκτική πολιτική φορολογική στα θέματα της φορολογίας. Υπάρχουν κάποιες ασυνέχειες και ασυνέπειες. Για παράδειγμα, οι περισσότερες χώρες της Ένωσης ε, δεν μπορούν να βρουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη μιας εταιρείας και γι' αυτό θα έπρεπε να επεκτείνουμε την υποχρέωση και την νομοθεσία σε όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. Κάποια νέα στοιχεία, τα οποία θεωρώ τα χρήσιμα, έχουν να κάνουν με, το λεγόμενο, με τη λεγόμενη μαύρη λίστα των φορολογικών παραδείσων. Υπάρχει μια λίστα του ΟΣΑ αυτή τη στιγμή, ίσως να μην είναι η πληρέστερη, γι' αυτό και καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτήσει ένα δικό του κατάλογο φορολογικών παραδείσων, μια νέα μαύρη λίστα. Αυτή είναι μια πρόταση που θα διατυπώσουμε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω τη σημασία της πρόταση της Ellis Line τα Ηνωμένα Έθνη να καταστούν ένας κομβικός παράγοντας. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι έγκαιρη η πρόταση και πάρα πολύ εύστοχη η πρόταση που λέει ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα έπρεπε να καταρτήσουν ένα φορολογική σύμβαση και να έχουν και ένα φορέα που ασχολείται με διεθνή φορολογικά ζητήματα. Η Νορβηγία, από ό,τι γνωρίζω, δραστηριοποιείται και αναζητεί υποστήριξη για να υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία υπό το ΝΟΙΕ. Επίσης χαίρομαι που στο σχέδιο έκθεσης αναφέρεται η ανάλυση με βάση το φύλλο και επειδή και εσείς είστε υπεύθυνοι για την περίληψη της διάστασης του φίλου σε όλες πολιτικές, είναι καλό και με την ίσπραξη εσόδων θα μπορούσε να, καταπολεμηθεί, να μπορούσαν να καταπολεμηθούν οι ανισότητες μεταξύ των δύο φίλων και να αυξηθούν οι δυνατότητες κοινωνικής προστασίας και ούτω καθεξής. Αυτά, κατά βάση μια πολύ καλή πρόταση, θα συνεργαστούμε μαζί σας κύριε Σλάιν για να έχουμε μια, μια έκθεση που θα επηρεάσει πραγματικά τη δράση της Ένωσης στον κόσμο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Νάτσιο Κοράο καταρχάς και με τον κ. Σίλα Περέιρα. Ευχαριστώ. Πιστεύω πως ε, η βασική εργασία της Ελισβάνη είναι εξαιρετική. Εξάλλου είναι συμπληρωματική στην έκθεση του Σίλβα Περέιρα για την διάσκεψη της Αντισαμπέμπα και άρα την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Και είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σημαντικό οι δύο αυτές εκθέσεις να συμβαδίσουν. Τα σημεία που απαριθμόνται είναι, είμαι σύμφωνος και, μάλλον και το θέμα ε, είναι εκείνο ε, που αφορά τι αναπτυσσόμενε χώρε που είναι με φορολογική παράδειση. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και είναι δύσκολο στην επίλυσή του, γιατί ο συνάδελφο αναφέρθηκε ακριβώ στο γεγονό ότι συχνά δεν καταφέρνουν να πληρώνουν τους φόρους σε ένα συγκεκριμένο μέρος γιατί ε, μεταφέρονται τα κεφάλαια σε άλλες χώρες. Στην πραγματικότητα γίνεται μόνο και μόνο λόγω ενός, ε, λόγω ε, φορολογικού shopping επιλογής, ε, δηλαδή που ισχύουν οι καλύτερε Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο πολύ ε, ε, εφάνταστα έχει οικοδομηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο εάν, εφόσον είναι φιλελεύθερες πολιτικές που κυβερνούν τον κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κατάλληλα μέσα ώστε να βρούμε λύσεις. Σίγουρα στη διάρκεια των συνεδριάσεων ανάμεσα στον ε, εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές θα μπορέσουμε να βρούμε κάτι πιο αποτελεσματικό. Κατά τα λοιπά, θεωρώ πως το ε, σχέδιο είναι καλό. Τα σημεία και οι παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί είναι θετικές και με βρίσκουν σύμφωνα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Περέιρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ παίρνω το λόγο για να συγχαρώ την εισηγήτρια Έλλης Λάινε για την εξαιρετική έκθεση που μας παρουσίασε και επίσης για να επιβεβαιώσω ότι η έκθεση αυτή συμβαδίζει με το βασικό νόημα της δικής μου έκθεσης σε σχέση με τη διάσκεψη της Αντισαμπέμπα και της χρηματοδότησης της ανάπτυξης μετά το 2015 και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ένας από τους βασικούς, τις βασικές στοιχές μιας σημαντικής ατζέντα για την αναπτυξιακή βοήθεια και τη δυνατότητα κινητοποίησης των εγχώριων πόρων αλλά και η βελτίωση των φορολογικών συστημάτων ώστε να είναι αποτελεσματικά και δίκαια αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει όντω να γίνει η χρήση και κινητοποίηση όλων αυτών των πόρων. Και όταν βλέπουμε ότι κάποιοι εκφράζουν ανησυχίε για το θέμα της ε, διαφθορά, που είναι πραγματικό στις αναπτυσσόμενε χώρες, αυτό είναι το κεφάλαιο όπου ε, η κατάσταση δεν έχει μεγάλο πολύ νόημα γιατί κάποιες φορέ φαίνεται να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι επειδή υπάρχει ε, διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, θα είναι ε, μάταιο το να επενδύσουμε στα φορολογικά συστήματα ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η διαφθορά. Είναι ακριβώ το αντίθετο που ισχύει. Ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα το οποίο είναι καλά ενσωματωμένο διεθνώ σε συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών πιο αποτελεσματικό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την διαφθορά στι αναπτυσσόμενε χώρε. Θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω μια πρόταση ε, που υπάρχει στην ε, έκθεση Line και είναι και στη δική μου έκθεση και είναι η ιδέα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργηθεί ένα όργανο με τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να συζητηθεί η, διεθνή διεθνής φορολογική συνεργασία. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να ε, υποστηρίζουμε ότι η διεθνής φορολογική συνεργασία είναι ένα σύνολο υποδείξεων που απευθύνουν οι αναπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες. Πρέπει να συμμετέχουν στη συζήτηση για τους κανόνες συνεργασίας σε θέματα φορολογικά και αυτό δεν μπορούσε να γίνει νομίζω πιο κατά, σωστά στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Και εγώ να πω ότι συμφωνώ με τον Πέντρο Σίλβα Περέιρα. πρέπει να δράσουμε ε, για αυτό το θέμα των φόρων για να δούμε πού καταβάλλονται οι φόροι. Έχουμε και εμείς θέματα φορολογικά. Δεν τα έχουν τα προβλήματα μόνο οι αναπτυσσόμενες χώρες. Βλέπουμε εταιρείε που προσπαθούν να αποφύγουν διαρκώς πώς να πληρώσουν φόρους, αλλά αν δεν έχουμε φόρους δεν μπορούμε να έχουμε την κοινωνία που θέλουμε. Χρειάζεται λοιπόν δράση και πρέπει να είναι διεθνή η δράση για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο που δεν είναι ίδιον των αναπτυσσόμενων χωρών. Βλέπουμε και εδώ διαρκώς φορολογικά σκάνδαλα που ξεσπάνε στην Ένωση. Και γι' αυτό και οι πολίτες μας χάνουν την πίστη του, γιατί αισθάνονται ότι αυτοί ε, επιβαρύνονται, ενώ οι εταιρείε όχι. Δεν είναι θέμα δεξιάς-αριστεράς, είναι ένα πρόβλημα το με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί κάθε κόμμα. Δεν έχω κάποιον από την Κομισιόν. Α, ε, ε, θέλετε κάτι να μας πείτε σύντομα παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την έκθεση. Είναι μια εξαιρετική έκθεση. Συμφωνούμε απόλυτα τα αρνητικά, στις αρνητικές επιπτώσεις της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής στι ε, στις χώρε και πρέπει να όντως να αναπτυχθούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, να υπάρχουν ισότιμοι όροι οικονομική ε, ολοκλήρωση σημαίνει πως αυτά τα πράγματα θα πρέπει να εξεταστούν σε παγκόσμιο επίπεδο και βέβαια η κινητοποίηση χώρη και η καταπολέμηση των παράνομων ε, ε, οικονομικών ροών είναι ένα σημαντικό τμήμα ένα σημαντικό θέμα μάλλον για την Αντίσα αλλά και για την διαπραγματεύση μετά το 2015. Η Κομισιόν είναι βασικός παίκτη Έχουμε πιέσει στην ε, ομάδα των G20 αλλά και στον ΩΣΑ για να βελτιωθεί το πρόγραμμα δράσης PAPS. Ε, έχουμε διαρκώς τονίσει την στήριξή μας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες σε επίπεδο χώρας, περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο πιέζουμε ώστε να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ε, ικανότητες μέσα στο φορολογικό σύστημα, ώστε να μπορούν όχι μόνο να, να κάνουν σωστή ε, δημοσιονομική διαχείριση, αλλά και να κατοπολεμήσουν τις παράνομες δημοσιονομικές ροές και βέβαια τη φοροδιαφυγή. Θα φτιάξουμε ένα έγγραφο εργασίας, ίσως όχι ανακοίνωση, ε, για την φορολογία και την ανάπτυξη, γιατί πιστεύουμε ότι η ανακοίνωση του 2010 εξακολουθεί να είναι έγκυρη και να ισχύει. Επίσης κάποιος μίλησε για τα χρήματα και το στόμα, κάτι τέτοιο. Εμείς ε, θα υποβάλουμε πρωτοβουλία όσον αφορά το θεματικό πρόγραμμα για τα παγκόσμια δημόσια αγαθά. Α, συγγνώμη, δεν σας ρώτησα πώς σας λένε, μπορείτε να μας πείτε. Να ξέρουμε με ποιον συνομιλούμε. πολύ συχνά στη χώρα μου μιλάμε για πρόσωπους γραφειοκράτες. Ονομάζομαι Σούσαν Βίλερ, είμαι να αναπληρωματική κόστιματάρχη της μονάδας ε, για τη δημόσια ε, διαχείριση στην ΤΕΦΚΟ. Ε, ο τμηματάρχης μας είναι ήδη διακοπές. εντάξει, επιτρέπεται. ναι, ειδικά για έναν άντρα που πάει διακοπές στα παιδιά του, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ρώτησα το όνομά σας γιατί μπορεί να θέλει να τους επαφή μαζί σας. κυρία Σλάιν, θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους για τα πολύτιμά σας σχόλια και τα σημείωσα όλα και θα με απασχολήσουν στη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που εν γέννη εκτιμήσατε τη δομή που σκέφτηκα να δώσω σε αυτή την ε, έκθεση. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε επί τη βάση των όσων είπαμε και σήμερα και ο ρόλος μου θα είναι να προσπαθήσω να βρω όσο γίνεται πιο σύντομα κοινέ θέσεις για αυτά τα σπουδαία ζητήματα και να προτείνω κοινέ λύσεις. Όπως είπατε πολύ, είναι απαραίτητο να έχουμε μια γενική οπτική σε αυτό το θέμα, γιατί είναι προφανές ότι ζούμε σε καιρούς όπου μπορούν να κινηθούν ε, τεράστια κεφάλαια ε, από τη μια μεριά στην άλλη του κόσμου με ένα κλικ. Ε, χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε πιο, σε πιο ψηλό επίπεδο για να βρούμε πιο κοινέ και αποτελεσματικές λύσεις. Ευχαριστώ όλος ιδιαίτερα τον Πέντρο για τη συμβολή του και για την έκθεσή του αλλά και για το, τις συνήξεις που μου έκανε σήμερα και ελπίζω πως θα συμμετέχει και στον περιττέρω προγραμματισμό και ευχαριστώ και την Κομισιόν για το πνεύμα συνεργασίας, ε, είναι θετική και για το διάλογο που θα έχουμε από τώρα μέχρι την ε, ψήφιση της έκθεσης μου. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω άλλο, γιατί ορισμένοι συνάδελφοι έχουν ήδη φύγει. Ανανεώνω τη βούλησή μου να συνεργαστώ με όλους και ελπίζω πως ε, σύντομα θα έχουμε την επόμενη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Έλλη. Να πω απλά ότι η προθέσμα κατάσταση τροπολογιών είναι η 30 Απριλίου στι 12 και θα ψηφίσουμε, μάλλον θα έχουμε ανταλλαγή ε, απόψεων 6 Μαΐου και 1 Ιουνίου θα ψηφίσουμε. Σίγουρα θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε έγκαιρα. Ελπίζουμε και το έγγραφο εργασία τη Κομισιόν και την συνεδρία τη Συναντήσα Μπέμπα. Και αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο σημαντικό σημείο τη μέσα διάταξη. υπάρχουν 18 ώρα των ερωτήσεων. Μαρία Χόλμπρουκ έχει μια ερώτηση η οποία αφορά την καλλιέργεια ζάχαρο, ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, ζαχαροκάλαμο τέλος πάντων. Και έχουμε και το θέμα της ε, ζαχαρότητας πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2005 είχε ε, ληφθεί μια απόφαση να πάψει το σύστημα των ποσοστώσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τότε είχαμε θεσπίσει ειδικά υποστηρικτικά μέτρα, ένα πρόγραμμα για τους καλλιεργητές αγροκάλαμου χώρες ΑΚΕ που ενδεχομένως επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές στην αγορά. Η Μαρία και άλλοι, και εγώ και άλλοι ακούσαμε ότι πλήττονται οι αγρότες, επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε την Κομισιόν καταρχάς και Μαρία μετά θα σου δώσω το λόγο. Η Κομισιόν. Ναι. Μάνφρεντ Μπραντ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Manfred Μπάντ λέγομαι, δουλεύω στην ΤΕΦΚΟ, είμαι Γενικός Διευθυντής Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης στη ΣΥΕΝΑ, μάλλον στη Γενική Διεύθυνση, ε, είμαι στην ομάδα, μονάδα ΣΥΕΝΑ, ο προϊστάμενος μου είναι διακοπές και στα συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα και και καταρχάς να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμερίζεται απόλυτα την άποψη ότι οι συνοδευτικά μέτρα για τις χώρες του πρωτοκόλλου ζάχαρης ε, δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής επαρκώς ε, στις ε, ανάγκες των πληγισών κοινοτήτων. Το 2006 οι χώρες του πρωτοκόλλου ζάχαρης έλαβαν 1,2 δις ευρώ για υπομορφή βοήθειας αναδιάρθρωσης και συνοδευτικών μέτρων για αυτές τις χώρες πρωτοκόλλου ζάχαρης, ένα πρόγραμμα που έδωσε ένα ευρύ πλαίσιο ε, μέτρων για αυτές τις χώρες, ε, ε, προετοιμαζόμενες όπως θα έπρεπε αυτές τις χώρες για τη λήξη του καθεστώτος στον τομέα του ζαχαροκάλαμου. Και επίσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφοροποίηση περιοχών εξαρτημένων από αυτή την καλλιέργεια και να βοηθήσει στην προσαρμογή. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι, χώρες, οι δικαιούχες χώρες δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν όλα τα κονδύλια τους διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούν να υπάρχουν προγράμματα ε, και 340 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν ε, αδιάθετα. Και Γι' αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο ε, πρέπει να. Μάλλον πρέπει να γίνουν σημαντικότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά την βοήθεια και την, το μετρησμό της φτώχεια, έχουμε το 11ο ΕΤΑ 30,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν για τις χώρες ΑΚΕ. Τα περισσότερα πολιετή ενδεικτικά προγράμματα έχουν υπογραφεί, καταρτίστηκαν αυτά τα προγράμματα, συμφωνήθηκαν με συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, εθνικών αρχών, κοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται για κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τη βιώσιμη μείωση τη στόχη και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για μέτρα αναδιάρθρωση για όσου ε, αγρότε δεν μπορούν να προσαρμοστούν στι ε, εξελίξει τη αγορά. Οι πολιτικέ επιλογέ ουσιαστικά είναι στα χέρια των χωρών εταίρων και των εμπλεκομένων μερών που είναι και αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις η ζάχαρη είχε επιλογή ως υποσχόμενος πολλά, πολλά υποσχόμενος για ανάπτυξη απασχόληση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ανάλυση και οι επιλογές κατέληξαν ότι πρέπει να γίνει στροφή σε άλλες δραστηριότητες και σε άλλους τομείς. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τη δήλωσή σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει μικρές εκμεταλλεύσεις από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και χώρες ΑΚΕ να εξάγουν ε, ε, ζάχαρη από ζαχαροκάλυμο. Αυτό δεν είναι σωστό διότι αυτά προγραμματίζονται, αποφασίζονται αναπερίπτωση. Αυτά ήθελα να πω και να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου την Γάμα Δέλτα Γεωργία ο οποίος θα σας απαντήσει πάνω σε κάποιες άλλες πτυχές αυτών των ερωτήσεων. Thank I'm Jules from Jules Δέλτα Άγκρι από τη μονάδα Α3 και είμαι αρμόδιος για τις χώρες ΑΚΕ και τα αναπτυξιακά ζητήματα και ο δικός μου προϊστάμενος ε, απουσιάζει, θα λάβω λοιπόν εγώ το λόγο, αν μου επιτρέπετε. Σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν περιλάμβανε καμία αλλαγή στο εμπορικό καθεστώς ε, και στην προτιμησιακή πρόσβαση για τους ε, προμηθευτές ε, ζάχαρης της χώρας και δεν είναι μια νέα ιδέα η κατάσταση των ποσοστώσεων. Είχαμε ήδη το 2006 μετάρρυθμιση της ΚΟΑ ζάχαρης και είχε εκεί φανεί ότι μέχρι το 2013 ή μάλλον 2015 το εμπορία θα σταματούσε χωρίς ποσόστοση. Αποφασίστηκε παρόλα αυτά να επεκταθεί αυτό το καθεστώ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 και εκεί να σταματήσουν οι ποσοστώσει ζάχαρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρίσμα της ε, τρέχουσας κατάστασης ε, και το που πηγαίνει η ΚΑΠ με την προσανατοσμό των αγορών, η κατάργηση των ποσοστώσεων είναι αναπόφευκτη γιατί δημιουργεί ακαμψίες και δεν επιτρέπει στην βιομηχανία της ζάχαρης να ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές αγοράς. Κατάργηση ε, της ποσότητας παραγωγής ζάχαρης θα πρέπει να ερμηνευθεί ε, με τα εξή υπόψη. Πρώτον, η πρόταση δεν αλλάζει τις εμπορικές διευθετήσεις για τη ζάχαρη. Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με χώρες ΑΚΕ με λιγότερο ε, αναπτυγμένες χώρες παραμένουν, άρα αυτές οι χώρες θα παραμείνουν οι δικαιούχοι αυτής της προτιμησιακής αδοσμολόγητης ε, πρόσβασης. Έχουμε το, Γιαουντέ, το Λομέ και το Κοτονού. δεν οδήγησαν αυτές οι συνθήκες σε διαφοροποίηση των οικονομιών. Γι' αυτό θελήσαμε να έχουμε ασύμετρες ε, οικονομικέ ε, οικονομικές εταιρικές σχέσεις ε, με μονομένες χώρες ε, για τα τυπάσματα, τα μηχανήματα, τους πόρους, ώστε να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και βέβαια παρέχεται και ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές της Ένωσης. Δεύτερον, θα χρειαστούν εισαγωγέ για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μας επειδή έχουμε και πολλά εργοστάσια ευγενισμού ζάχαρης, άρα χρειαζόμαστε εισαγωγέ πρώτης ύλη ζάχαρης. Επίσης θα σας πω ότι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για το μέλλον της αγοράς της ζάχαρης εγκροτήθηκε πολύ πρόσφατα και θα παρακολουθεί την κατάσταση της αγοράς, τα στατιστικά στοιχεία, τις τιμές και το πώς επηρεάζει η πρόταση η μεταρρυθμιστική. Ε, την κατάσταση. Αναλύουμε λοιπόν όλα αυτά, αναλύουμε και τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων στις χώρες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προσκληθεί ως, ε, όπως και όλοι σε άλλες ομάδες, όπως και σε όλες τις άλλες ομάδες εμπειρογνωμών και σε αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Μπορούμε να σας δώσουμε άλλες πληροφορίες, αν θέλετε, για τον πρώτο εργασιών αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ τώρα, κυρία Χούντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι ότι οι εμπορικές συμφωνίες αυτές δεν άλλαξαν και η πρόσβαση στην αγορά παραμένει ίδια. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι η τιμή της ζάχαρης τα τελευταία χρόνια διακινδυνεύει και υπονομεύει τις μικρές επιχειρήσεις ε, στις χώρες ΑΚΕ. Και κλείνει το μικρόφωνο της ομιλητρίας. Oh, sorry. Und es ist immer noch. Και η διαφοροποίηση στις χώρες αυτές έχει παρουσιαστεί με λυπή τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να εξετάσουμε τις ποσοστώσεις ζάχαρης και να δούμε πώς η εμπλεκόμενες χώρες. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στις εμπλεκόμενες χώρες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα πρέπει να ελέγχουμε με συνεχτικό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εμπορικές μας συμφωνίες και συμβάσεις. Παράλληλα καταπολεμώντας σε παγκόσμιο επίπεδο τη φτώχεια. Καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή κάνει προσπάθειες για τη σάχαρη, αλλά να συνειδητοποιούμε το τι συμβαίνει και στις χώρες. Πολύ απλά δεν, φτάνει, δεν φτάνουν αυτά που γίνονται για να προστατευτεί το βιός και οι επιχειρήσει των μικρομεσαίων. Η πρόεδρος δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις όμως. Θυμάμαι την μεταρρύθμιση της ζάχαρης, αυτά που έγινε το 2006, γιατί ήμουν ένα αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής αυτής και ήταν εδώ η Γκλένης Κένετ και συζητήσαμε τα σχετικά μέτρα. και τα μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τους αγρότες. Αναρωτιέμαι όμως αν έχει, γίνεται, αν έχει γίνει ανάλυση για τον αντίκτυπο των όσων έγιναν και το τι έγινε πραγματικά για να βοηθηθούν οι αγρότες η παραγωγή ζαχαροκαλαμού. Υπήρξαν μέτρα, αλλά τα μέτρα αυτά έδωσαν τροφή στους ε, αγρότες. Και ποιος ωφελήθηκε από τη μεταρρύθμιση τελικά, γιατί τότε μας είχαν πει ότι θα μειωθούν οι τιμές για τον καταναλωτή, θα πέσουν και θα σταματήσουν, θα καταργηθούν και οι ποσοστώσεις για το γάλα και τελικά Ποιο ωφελήθηκε, ο καταναλωτή ή οι μεγάλε εταιρείε. Άλλα μας λένε όμως οι ακρότες επιτόπου δεν νιώθουν ότι τους υποθερήξαμε να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους. Εσείς λοιπόν τι διαπιστώνετε και ίσως ε, πριν ε, είναι πολύ αργά μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε την πολιτική αυτή για να δούμε κατά πόσο λειτουργεί. Γιατί εσείς μας λέτε ότι έχουμε λεφτά και ότι συνέβησαν όλα αυτά, αλλά δεν μας δεν συνάδουν αυτά με αυτά που μας λέει και ο κόσμος. Ποιος ευφυλήθηκε λοιπόν από τη μεταρρύθμιση. Ίσως και συνάδελφοι από τα γεωργικά θέματα θα μπορούσαν να μας πούν τι γίνεται κατά πόσον υπάρχει υποστήριξη της παραγωγής. γιατί κάποιες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο υποστήριξη των παραγωγών σαχαροκάλαμου. Αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ή μήπως αυτό θα φέρει ακόμα σε πιο δύσκολη θέση τον ανταγωνισμό με τους αγρότες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Χόεμπρούχου για τις ερωτήσεις αυτές. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και ύστερα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω από την τελευταία παρατήρηση που κάνατε. Ποιο ε, ωφελήθηκε από την μεταρρύθμιση, έγινε η διάμεση να θεώρηση το 2010. Δεν ήταν καθοριστική. Έχουμε ακόμα 17 προγράμματα που είναι ακόμα λειτουργικά. 340 εκατομμύρια ευρώ να τα απαντηθούν ακόμα. Ως συνήθως, υποθέτω, δεν έχω επιβέωση από την υπηρεσία αξιολόγησης, αλλά μέτρα από το MSSP αξιολογηθούν για το κατά πόσο ήταν αποτελεσματικά. Για ποιον ωφέλησαν. Είναι δύσκολο να κάνουμε τώρα μια δήλωση δεσμευτική γιατί το πρόγραμμα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διορίσει εξωτερικού ε, αξιολογητέ για να είναι αντικειμενική η αξιολόγηση. Είναι πρόωρο. Τώρα το με αυτό. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ακόμα. Είμαι βέβαιο ότι θα γίνει μια τελική αξιολόγηση του χρόνου ή σε δύο χρόνια όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πλειονότητα των προγραμμάτων. Όπως τόνισα όμως προσπαθούμε να γίνεται προγραμματισμός μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό αποτελεί πάντα κοινή πρακτική. Για το ερώτημα τώρα και τα σχόλια της κυρία Χόιμπρου. Αναφερθήκατε και υπογραμμίσατε ότι η τιμή της σάχαρης δραστικά μειώθηκε. Και μάλιστα σε ένα επίπεδο όπου είναι πολύ δύσκολο για τον παραγωγό να επιβιώσει με την παραγωγή σαχαροκόλαμου. Το 2006, όταν ξεκίνησε το μέτριο, ήταν σαφές ότι ήταν τεχνητά υψηλέ οι τιμέ και μη βιώσιμα υψηλέ μάλιστα. Αυτό ήταν και ο σκοπό του μέτρου. Αν θέλουμε να υπάρχει ανταγωνιστικό πλανέκτημα για την παραγωγή ζαχαροκάλαμου, θα πρέπει να γίνεται η παραγωγή πιο αποτελεσματική για να καταστρέψουμε τη σειρά της πιο ανταγωνιστική όπου μακροπρόθεσμα δεν έχει νόημα οι χώρες λόγω των εδαφικών συνθήκων, λόγω των υπόλοιπων συνθήκων δεν είναι σε θέση Ήταν από τότε σαφέ δηλαδή ότι η τιμή λίγο πολύ θα σταθεροποιούταν και θα έπρεπε στα 300 ευρώ ανά τόνο. Αν λοιπόν δεν είναι ανταγωνιστική η παραγωγή, θα έπρεπε να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους οι αγρότες. Αυτό ήταν σαφώς ένας από τους στόχους του EMSP. Γιατί δεν συνέβη τώρα αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Όντως, αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί στην τελική αξιολόγηση, αλλά εγώ προσωπικά φαντάζομαι ότι το γεγονός ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι λόγω των πλεονεκτημάτων που είχαν ε, οι αγρότες αυτοί τεχνητά προτιμούσαν να μην προβούν σε διαφοροποίηση. Εμείς ε, παρόλα αυτά προσπαθήσαμε να πετύχουμε την διαφοροποίηση σε μέρη όπου δεν υπήρχε συγκριτικό πλεονέκτημα. Τώρα το κατά πόσο το πετύχαμε και στι περιπτώσει που το πετύχαμε, ποιος έφταγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι σε στόχο. Δεν ξέρω αυτό, θα δούμε. Αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο σε πρώτη φάση. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Το επίπεδο τιμών που διαπιστώθηκε το 2012-2013 700 ευρώ και πάνω ανατόνο δεν ήταν βιώσιμο ήταν διπλάσιο και παραπάνω από τις κανονικές τιμές. Οι τιμές λοιπόν έπεσαν στα 433 ευρώ ανατόνο για τη λευκή ζάχαρη. Αλλά εξακολουθούν να είναι 100 ευρώ παραπάνω ανατόνο δεν υπήρξε αντίκτυπο ε, στην παγκόσμια αγορά λόγω του συστήματος προσωστώσεων το 2017. Η ζάχαρη για τους ε, Βραζιλιάνους εξαγωγούς είναι πολύ ελκυστικό προϊόν και ο ενδικός η ειδική παραγωγή είναι μεγαλύτερη και όλο και πιο πολλές ε, εξαγωγές βλέπουμε και επιδοτήσει των εξαγωγών. Ρωτήσατε κατά πόσον η άμεση αρρωγή μπορεί να βοηθήσει την παραγωγή. Ναι, 10 κράτη-μέλη αναφέραν ότι θα εφάρμοζαν το μέτρο στο, στον τομέα του ζαχαρόταστου του ζαχαρότευλου για την άμεση βοήθεια. Αλλά τέτοιου είδους υποστηρίξη δεν έχει σκοπό να αυξήσει την παραγωγή. Ισχύει μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένε ανάγκες. Και η ομάδα για τη ζάχαρη στην Ευρώπη που συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και συνεδρίασε. Διαπίστωσα ότι το μερίδιο της ομάδας αυτής είναι 4% της άμεσης υποστήριξης. Και προφανώς, αν θέλετε, μπορώ να δώσουμε πιο πολλέ πληροφορίε. Και θα υπάρξει από ό,τι κατάλαβα και η ειδική συνεδρία τη Επιτροπής ε, Γεωργικών Υποθέσεων για το θέμα τη ζάχαρης. Να προσθέσω τέλος τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξη για την εξέλιξη της αγορά τη ζάχαρης οι αναπτυσσόμενες αγορές δεν υπονομεύονται, δεν, διακυβεύονται. Ξέρουμε όμως ότι θα μειωθούν σε κάποιο βαθμό οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Μία ερώτηση να κάνω. Τι χρήματα εκπροσωπεί αυτό το 4%, αντιπροσωπεύει αυτό το 4% της άμεσης υποστήριξης, γιατί κλίμακα κονδυλίων μιλάμε. Ναι, ακούστε, μιλάμε για, για, για, για, για, 176 εκατομμύρια. 176 εκατομμύρια, μάλιστα, λέει πρόεδρος. Τέλος. Τον σάφω από την ΤΕΦΚΟ. Είπατε θα κάνετε την επιστολή μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν είναι λίγο αργά. Να περιμένουμε δύο χρόνια ακόμη να λήξει το πρόγραμμα και να εξολογήσουμε και να δούμε πήγαν ή δεν πήγαν τα χρήματα στους ε, αγρότες και μετά να κλαίμε γιατί δεν τα πήρανε και ήταν αντιπαραγωγικό. Έχετε ε, κάποιες ε, αντιπροσωπείες στις χώρες και αυτές λαμβάνουν αποφάσεις, έτσι δεν είναι. Μπορείτε να ρωτήσετε τις αντιπροσωπείες την επόμενη εβδομάδα. Τι κάνουνε, πάνε τα χρήματα στους ε, αγρότες. Καταλαβαίνω το θέμα των εταιρικών σχέσεων με άλλες χώρες, θα ήταν όμως εμείς να ξέρουμε νωρίτερα και όχι να καθόμαστε και να περιμένουμε δύο χρόνια και να πούμε μετά «Α, τι κρίμα, αλλά έγινε» και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αφού έχουμε 340 εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουμε προγραμματίσει που θα τα βάλουμε, μήπως με τις αντιπροσωπείες έχουμε μια τύχη και μια ευκαιρία να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα αν δεν λειτουργούν τώρα καλά. Απάντηση. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μιλάμε για 1,2 δις τα οποία δαπανήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια σε 18 διαφορετικές χώρες. Γι' αυτό είπα αξιολόγηση, αναφερόμουν βέβαια στη συνολική αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος. Είναι κοινή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνεται και μια ενδιάμεση αξιολόγηση πάντοτε, οπότε επαναπροσανατολίζουμε, ανακατευθύνουμε το πρόγραμμα αν χρειάζεται, γιατί όπως πολύ σωστά είπα τέλος δεν έχει νόημα και μετά έχουμε την τελική αξιολόγηση. Επί προσθέτως, αλλά σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν έχω στη θέση μου αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Επιπροσθέτως, η συνήθω πρακτική, εγώ ξέρετε έχω εργαστεί σε πέντε διαφορετικές αντιπροσωπείες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας το λέω ειλικρινά, ποτέ δεν είδα να έχουμε ένα πρόγραμμα, πόσο μάλλον ευαίσθητο λεπτό πρόγραμμα που είναι η ζάχαρη, ένα ευαίσθητο προϊόν, ιδίω αν εργάζεται κανεί ε, ε για μια, ένα προσαλισμό τη πολιτική. Σε αυτή την ε, αξιολόγηση που γίνεται ενδιάμεσα και τελικά γίνεται ειδικά για το κάθε πρόγραμμα. Όταν έχουμε ένα ευαίσθητο πρόγραμμα μάλιστα, πολλές φορές κάνουμε δύο ενδιάμεσα αξιολόγηση. Τη μία την κάνουμε αρκετά νωρίς, ένα χρόνο ε, αφού ξεκίνησε. Έχουμε τη μελέτη της σκοπιμότητας η οποία εξετάζει τις λεπτομέρειες του προγραμματισμού και όταν είναι ένα ευαίσθητο πρόγραμμα ένα χρόνο μετά την έναρξή του γίνεται η πρώτη διάμεση, μετά γίνεται η δεύτερη διάμεση αξιολόγηση, έτσι ώστε να γίνουν οι κρίσιμε παρατηρήσεις. Αν κάτι έχει βγει εκτό τροχιάς, να μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα. Αυτή είναι η δική μου προσωπική εμπειρία. Ήμουν και στη Γουιάννα, ξέρετε, που είναι ε, παραγωγός ζάχαρης. Ε, αυτή ήταν η κοινή πρακτική. Όταν μίλησα λοιπόν για αξιολόγηση, αναφέρθηκα μόνο στην αξιολόγηση όλου του προγράμματος συνολικά. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτοί που μας είπαν ότι υπάρχουν πρόβλημα, ίσως να μας πούνε παραπάνω πράγματα και θα επανέλθω. Α, ναι, μου επιτρέπετε να διευκρινίσω κι εγώ κάτι. Αυτό το 4% δεν έχει να κάνει με το σύνολο, αλλά με το 4% της ε, προβλεπόμενης ε, συνδεδεμένης ε, στήριξης. Well, can I thank you very much for... Uh, can I thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα επανέλθουμε, όπως σας είπα, σε σημείο 19 διάφορα. Έχουμε τίποτα, όχι. Επόμενη συνεδρίαση. 20 Απριλίου στις 3 το μεσημέρι. Τελειώνουμε λίγο νωρίτερα, καλό αυτό, γιατί ξεκινάνε απόψε διακοπές. Ε, σε όσους συναδέλφου ε, θα γυρίσουν στις ώρες τους, εύχομαι καλή επιστροφή. Και όσοι πάνε διακοπές, ε, καλό Σαββατοκύριακο, καλό Πάσχα. Ευχαριστή και τους διερμηνείς που τόσες φορές μας έχουν παραχωρήσει έξτρα χρόνο. Τώρα φεύγουν λίγο νωρίτερα και αυτοί. Ευχαριστούμε.